Καλημέρα σα, ε, κύριε και κύριοι. Ξεκινήσουμε. Το πρώτο θέμα είναι η έγκριση τη μερίσιας διάταξης. Δεν ξέρω αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, να αλλάξουμε κάτι στη μερίσια διάταξη. Αν όχι, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Πάμε στο σημείο υπαρθμών 2, έγκριση των πρακτικών της ε, συνεδρίασης. Ε, το σχέδιο των πρακτικών της συνεδρίασης της 23-24 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου του 2019 ε, τα πρακτικά αυτά τα έχετε στο φάκελό σας και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, τα πρακτικά εγκρίνονται. Οι αντιρρήσεις βεβαίω μπορούν να καταθεθούν και μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Σημείο υπεριθμών 3 αποφάσεις των συντονιστών. Και εδώ ισχύει η ίδια διαδικασία. Έχουμε τις αποφάσεις των συντονιστών που ελήφθησαν στις 23 Σεπτεμβρίου και 2 Οκτωβρίου και αυτές συμπεριλαμβάνονται στα πρακτικά της συνεδρίασης. Και πάλι, εάν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης δεν κατατεθούν αντιρρήσεις και αυτά τα πρακτικά, οι αποφάσεις θα θεωρηθούν εγκεκριμένες. Σημείο υπερθμών 4. Η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Ε, μπορούμε να χαιρετήσουμε ανθρώπους από το Τελίνο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, στη Λισαβόνα, σε όλα τα μέρη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και διερμηνία. Παρακαλώ να μιλάτε ε, καθαρά, ε, αργά και καθαρά, για να γίνεται και σωστή διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Σημείο υπερθμών 5. Πρόκειται για την ε, σύναψη της συμφωνίας, τα συμπεράσματα με τη συμφωνία με την Ουκρανία, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία. το θέμα που διακυβεύεται είναι να έχουν οι Ουκρανοί μεγαλύτερες ποσοστώσεις για το κρέας πουλερικών που εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό εγκρίθηκε την προηγούμενη χρονιά, το Μάρτιο, τον Ιούλιο, ε, πήξαν περιττέρα ε, εξελίξεις. Η συγγήτριά μας είναι η κυρία Νίκο Γκιόρη και της δίνω το λόγο. Ε, καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα. Παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είπατε περί τίνος πρόκειται. Ε, στη συνεδρίασή μας συζητήσαμε γι' αυτό, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Κατ' ουσίαν πρόκειται για το εξής. Πρόκειται για ένα μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το φιλέτο κρέατος ε, από την Ουκρανία μπορεί να εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο με πολύ αυστηρές ε, προϋποθέσεις. Νομίζω αυτό αναφέρεται και στη συμφωνία. Τώρα, εκείνο το οποίο δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε, να προβλέψει ο νομοθέτης, είναι ότι θα εξακολουθεί να υπάρχει ένα παραθυράκι. Οι Ουκρανοί είναι ε, ευρηματικοί και βρήκαν αυτό το παραθυράκι ε, πρόκειται για καινοτόμους μεθόδους κοπής για να παρακάμπτονται οι ποσοστώσεις. Είναι περίφημη ε, ποικιλία Batman, δηλαδή κόβουν το φιλέτο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε στο φιλέτο περιλαμβάνεται και ένα μικρό ποδαράκι του κοτόπουλου και στην περίπτωση αυτή το κρέας αυτό μπορεί να εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χωρίς δασμούς. Κατ' ουσίαν δηλαδή ε, με, αυτή την, ε, με αυτό το τρίκ μπόρεσαν να βρουν μια λύση και με τον τρόπο αυτό ε, εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 55.000 τόνοι. Στην Ουκρανία είπαν ότι αυτό γίνεται, ότι γιατί όχι. Ε, βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τους Ουκρανούς και αυτό οδήγησε στο ότι τις ποσοστώσεις ε, συμπεριλαμβάνονται και δύο προστίκες. Πράγματι διατηρείται η ποσόστοση ε, και καταβάλλονται προσπάθειες να αποφευθεί αυτή η στρέβλωση της ε, αγοράς. Αυτό το θέμα απασχόλησε τους συναδέλφους στην Επιτροπή Γεωργίας. Υπάρχουν διατάξεις που αφορούν θέματα υγείας αυτές οι διατάξεις ε, ε, δεν ε, άλλαξαν και θα ήθελα λοιπόν να απευθυνθώ στην τους Ουκρανούς και να τους πω να σεβαστούν αυτή τη συμφωνία. Να μην ε, καταφεύγουν ε, σε ε, τρίκ και σε παραθυράκια. Το θέμα είναι πώς έχουμε προχωρήσει με αυτή τη συμφωνία. Σήμερα το πρωί έχω φρέσκες ειδήσει. Η Ουκρανική κυβέρνηση δέχτηκε αυτή τη συμφωνία και σήμερα το πρωί ε, μας δόθηκε η πληροφορία ότι αυτή η συμφωνία κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο προς ε, επικύρωση. Βεβαίως, Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι όταν το όλο θέμα θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο, θα σας ενημερώσω. Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν ότι παρακαλώ την Ουκρανία να προχωρήσει το των δυνατών, να μην καταφεύγει σε παραθυράκια και ή δυνατόν να εφαρμόζει πιστά αυτά τα οποία περιλαμβάνει η συμφωνία. Και το δεύτερο, θα ήθελα να παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους για το κατά πόσον τηρείται η συμφωνία. Ε, πρέπει να ε, λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις. Αυτό που έχει σημασία είναι, όπως σας είπα, να μην παραμένουν κενά στην νομοθεσία. Βεβαίως ε, λειτουργούμε καλή την πίστη, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και το ίδιο ε, προσδοκούμε και από τους εταίρους μας ε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι το όλο θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή Γεωργίας στηρίζει αυτά που σας είπα. Αυτό που θέλω να πω στους συναδέλφους είναι ότι νομίζω εδώ υπάρχουν πολλά και σημαντικά θέματα που θα πρέπει να λάβουμε μας και νομίζω θα ήταν σημαντικό να γίνει μια συζήτηση για το θέμα στην Ολομέλεια. Το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη, αλλά η όλη διαδικασία είναι διαδικασία συνένεσης και θα ήθελα να παρακαλέσω τον Πρόεδρο να οργανώσει μια ε, μικρή συζήτηση στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε και τώρα εκ μέρου των ε, σοσιαλδημοκρατών ε, Μάρικ Μπέκε, αλλά δεν είναι ε, παρόν και γι' αυτό τον δίνω το λόγο στη συντονίστρια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, λυπάται ο συνεισηγητής, ο σκιώδης ηγητής που δεν μπόρεσε να παραστεί σήμερα, αλλά μου έχει διαβιβάσει τα σχόλιά του και θα ήθελα να σας τα διαβάσω. Η ομάδα μας θεωρεί ότι η Συμφωνία Σύνδεση με την Ουκρανία είναι εξαιρετικά σημαντική, είναι ζωτικό εργαλείο για την προώθηση του εξυγχρονισμού της Ουκρανίας, του εκδημοκρατισμού και την ε, ύπαρξη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ποσοστώσει εισαγωγή μα επιτρέπουν να διασφαλίζουμε την εσωτερική μα αγορά, αλλά να δίνουμε και ευκαιρίε στους εταίρου μα. Με αυτόν τον τρόπο δεν διαταράσσονται και οι οικονομίε μα. Όμω, υπάρχει αυτό το παραθυράκι με το κρέα των πουλερικών που εξάγεται από την Ουκρανία προ την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί δεσμού και αυτό προκαλεί πολύ σοβαρέ ανισορροπίε. Και ήταν τεράστιο πλήγμα για τους ε, κτηνοτρόφους Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειάστηκε άμεση δράση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα μας εκφράζει τη λύπη της, διότι μέρος των τροπολογιών περιλαμβάνει την αύξηση των ποσοστώσεων και αυτό θα έχει αντίκτυπο στο γεωργικό τομέα, στο κλάδο της κτηνοτροφίας. Ε, η τροποποιημένη δεσμολογική συμφωνία θα εξεταστεί και πιστεύουμε ότι πρέπει να μπορέσει να προσφέρει λύση σε αυτή την προβληματική κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, κατά την οποία το κρέας των πουλερικών μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χωρίς κανένα περιορισμό ποσοστώσεων. Λόγω ε, αυτού του κενού στη ρύθμιση και θα πρέπει να παρακολουθήσετε στενά την εφαρμογή του DSFTA, του Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου, Ελευθέρων Συναλλαγών και έτσι ώστε να εφαρμόζεται αυτή όχι μόνο στο γράμμα αλλά και στο πνεύμα της. Και συμφωνώ με τον εισηγητή, πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσέγγιση. Ας γίνει μια σύντομη συζήτηση στην Ολομέλεια για να μπορέσουμε να εκπέμψουμε αυτό το μήνυμα και στον υπόλοιπο κόσμο, για να ε, γνωρίσουν όλη την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ ο σκιώδης συγητής για το Renew. Σας δίνω, δίνω σε εσά το λόγο. Συμφωνώ, στηρίζουμε τον εισηγητή. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομη. Τέλεια. Ο κύριος Μποξουά για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση και θέλω επίσης να συγχαρώ την Επιτροπή γιατί είχε διαχειριστεί αυτή την υπόθεση με εξαιρετικό τρόπο. Το είπε και η εισηγήτρια πολύ σωστά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε την εφαρμογή, την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας με αυτό το θέμα της συζήτηση στην Ολομέλεια ή της συζήτηση γενικότερα για τις λοιπές διατυπώσεις των συμφωνιών, των άλλων συμφωνιών που έχουμε με άλλες χώρες. Τι ακριβώς συμβαίνει, ε, θα αποσυρθεί ε, το θέμα το ουκρανικό. Θα σας απαντήσω μετά, λέει ο, ο πρόεδρος, ο Χέλμουτ Σόλτς για την Κούρια. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης. Καταρχήν, ακολουθούμε την εισηγητρία στη γραμμή της. Να τονίσω όμως ιδιαιτέρως ότι πρέπει να εξετάσουμε το θέμα πιο σφαιρικά, να μην περιοριστούμε μόνο στο κρέας των πολερικών, διότι υπάρχει μια επικίνδυνη εξέλιξη στην αγροδιατροφική βιομηχανία στην Ουκρανία. Συχνά μιλούμε για τη μακροοικονομική αρρωγή και θέλουμε να ξεχωρίσουμε τους κλάδους των εμπορικών μας σχέσεων και να τους εξετάζουμε ξεχωριστά. Υπάρχει καταστρατήγηση όμως της υποχρέωσης να χρησιμοποιηθεί το έσοδο από την παραγωγή για τη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Γι' αυτό θέλω λοιπόν να στηρίξω την εξής ιδέα. Να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό, και να το εξετάσουμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες για το πώς λειτουργεί και ποιους σκοπούς έχει ο γενικότερος κλάδος της αγροδιατροφικής βιομηχανίας στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, πολύ ωραία. Και τώρα για τους πράσινους, παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσής της. Έχω τρία σύντομα ερωτήματα. Βεβαίως στηρίζουμε την προσπάθεια της Ουκρανίας να υλοποιήσει πλήρως την Συμφωνία Σύνδεσης. Όμως οι πρακτικές αυτές ωφελούν μόνο τους ολιγάρχες και τους μεγάλους ομίλους. Θα πρέπει να αναλάβουμε ισχυρή δράση. Τι σχεδιάζει η Επιτροπή για να αποκαταστήσει την κατάσταση και για να διασφαλίσει ότι παρεμφερείς περιπτώσεις δεν θα συμβαίνουν είτε σε αυτόν τον κλάδο είτε σε άλλους κλάδους στο μέλλον. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Ε, αποκαλύφθηκε η υπόθεση, η υπόθεση και υπήρξε συνενοχή με τις τελωνιακές αρχές των κρατών μελών, οι οποίες έχουν εκδώσει νομικώς δεσμευτικές αποφάσεις που νομιμοποιούν το παράνομο αυτό εμπόριο. Έχει υπάρξει επίπτωση για αυτούς, κυρώσεις. Και τρίτη ερώτηση, σε σχέση με το κεκτημένο Έχουμε ε, συγκεκριμένε αδειοδοτήσεις για την ελεύθερη ε, εξαγωγική δραστηριότητα όπου να υπάρχει διευκόλυση τελωνίων. Ε, έχουν, έχει χορηγηθεί αυτό το καθεστώς του οικονομικού εμπορευόμενου μετά από έλεγχο. Όμως υπάρχουν κενά και έχουν βρεθεί προβληματικές καταστάσεις. Έχετε πάρει αυτά τα μέτρα για να αποκαταστήσετε το πρόβλημα και να μην υπάρχουν πια κενά στην νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Στρέφουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σουζάνα Μαρτσουέλα, αν προφέρω σωστά το όνομά σα, από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργία. Θα μα ενημερώσετε σχετικά. Καλημέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί πολύ γρήγορα εξετάσατε τον φάκελο αυτό, πολύ γρήγορα δώσατε τη συγκατάθεσή σας στην συμφωνία και έτσι μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του γεωργικού και κτηνοτροφικού κλάδου. Η λύση που συμφωνήσαμε με τις Ουκρανικές Αρχές είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να δοθεί ένα κατόφλι στις ενδυνάμια περιόριστες εξαγωγές ε, τέτοιου είδου κρέατος πολυερικών από την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 50.000 τόνους και αυτό το νούμερο είναι σημαντικό και πολλοί είπαν, είπατε ότι είναι κάτω από τις 55.000 τόνους που εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018. Χωρίς όριο, η Ουκρανία μπορεί να αυξήσει τις εξαγωγές της μελλοντικά και να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2018. Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι αυτό πράγματι μπορεί να συμβεί. Και γρήγορα και φέτος. Μετά την επιβράθυνση το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2018 αυξάνουν οι εισαγωγές από τον Ιανουάριο του 2019 και έφτασαν στα επίπεδα ρεκόρ 754 τόνους μόνο το Μάιο. Ιούνιο-Ιούλιο 42.000 και τόνους ε, κρέατος πουλερικών με αυτή τη συγκεκριμένη κοπή με την οποία γίνεται αδεσμός. Αν δεν βάλουμε όριο, μπορούμε να φτάσουμε εύκολα στους 70-80.000 τόνους μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας υιοθέτησε τη συμφωνία αυτή στις 23 Οκτωβρίου. Το Ουκρανικό Κοινοβούλιο πρέπει να προχωρήσει στην κύρωση της συμφωνίας. Θα κάνουμε το παν για να πείσουμε την Ουκρανική πλευρά να προχωρήσει γρήγορα, να κυρώσει τη συμφωνία για να ισχύσει το συντομότερο δυνατό, γιατί οι εξαγωγέ αυξάνονται ραγδαία είναι έτοιμη να εφαρμοστεί, εφαρμοστεί η εφαρμοστική πράξη της Κομισιόν για την αύξηση της ποσόστεσης μόλις κυρώσει τη συμφωνία το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την, παρακολου... εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και άλλων ε, συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, ελευθέρου εμπορίου. Επειδή το ζήτημα είναι πήγον, ενθαρρύνουμε τη δική σας Επιτροπή να υιοθετήσει τη γνωμοδότηση αύριο και να προχωρήσει ε, με αυτή τη διαδικασία συγκατάθεσης. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Και εγώ ευχαριστώ. Να επανέλθω στο ερώτημα του κυρίου Σμπουρζουά και άλλων ε, συνεισκιωδών εισηγητών. Ποια μαθήματα, ποια διδάγματα αντλήσατε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε οι μελλοντικέ συμφωνίες να μην έχουν τέτοιου είδους παραθυράκια. Ποια. We have checked all... Ακούστε, ελέγξαμε όλες τις συμφωνίες. Ε? που έχουμε διαπραγματευτεί. Και σε καμία άλλη συμφωνία δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιου είδους πρόβλημα. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα το γεγονός και πάντα ελέγχουμε ώστε να μην επαναληφθεί. Λάβετε υπόψη όμως ότι ήταν δύσκολο να προβλεφθεί αυτό που συνέβη στην προκειμένη περίπτωση. Δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο για να δούμε τι μπορεί να συμβαίνει σε άλλα προϊόντα ή άλλες συμφωνίες. Δεν υπήρχαν εμπορικέ συναλλαγές όταν έγινε η αλλες συμφωνιες δεν υπηρχαν εμπορικες συναλλαγες οταν εγινε η πραγματευση της συμφωνίας και δεν ήταν εύκολο να προβλέψουμε ότι θα εφεύρει αυτό το νέο τρόπο κοπής η Ουκρανία για να έχει πρόσβαση στην αγορά μας με αυτόν τον τρόπο. Ε, πρέπει να σας πω ότι άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την απάντηση. Το θέμα είναι πώς πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κενά. Προφανώς ε, και ε, μπορούμε να δούμε το όλο θέμα, αλλά πώς εφαρμόζεται η συμφωνία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και αν δούμε την, ε, τα αγροεπιχειρηματικά στην Ουκρανία, πράγματι συμφωνώ και εγώ, έχουμε ολιγαρχικές δομές που το μόνο που κάνουν είναι να προσπορίζονται το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος ε, και με τον τρόπο αυτό η Ουκρανία είναι ο μεγαλύτερος ε, προμηθευτής αυγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά ε, πού ακριβώς και πώς μπορούμε να αποκλείσουμε να μην διακυβεύονται όχι μόνο στο εσωτερικό τα συμφέροντά μας, αλλά να μεριμνήσουμε έτσι ώστε και στην Ουκρανία τα προσποριζόμενα κέρδη να επανέρχονται στο κράτος και εκεί να χρησιμοποιούνται για την βελτίωση, βελτίωση της ε, οικονομικής και εργασιακής κατάστασης. Ε, την επόμενη εβδομάδα θα καταθέσουμε μια σχετική μελέτη. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να έρθουν να την παρακολουθήσουν για να μπορούμε να ρίξουμε και μια ματιά στο παρασκήνιο της ε, όλης υπόθεσης. Ναι, να δούμε και με τη συνθήκη αν μπορούμε να βοηθήσουμε να κλείσουμε αυτά τα παραθυράκια. Η συγγήτρια, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλα τα σχόλια, για τις ανησυχίες που εξέφρασαν. Το είπα και εγώ άλλωστε ότι μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από την υπόθεση αυτή, να είμαστε προσεκτικοί και περιμένω να δείξει ιδιαίτερη προσοχή η Κομισιόν στις μελλοντικές της ενέργειες. Για να το πω και ομά, απαντώντας ταυτόχρονα στο συνάδελφο από το ECR. Είτε προχωρούμε ως έχει τώρα με την στρέβλωση της αγοράς και με τις ε, όλο και περισσότερο ε, αυξαμένες ε, τέτοιες παράνομες αυτού αυτού περίεργου είδους τεμαχίου κρέατος πουλερικών ή περιμένουμε να υπάρξει πραγματική και πιστή εφαρμογή της συμφωνίας από την Ουκρανική πλευρά. Γιατί επειδή το ρωτήσατε είναι ένα παραθυράκι, είναι μια πολύ ευφύης λύση που βρήκανε, που δεν είναι και παράνομη με βάση τη συμφωνία. Άρα προς το δικό μας το συμφέρον είναι να επανέλθουμε στο σύστημα των ποσοστώσεων. Για το στήθος Κοτόπουλου, όπως και αν κόβεται, με όποιο τρόπο και αν τεμαχίζεται, που μπορεί να φτάνει στις αγορές μας. Ε, να μην υπάρχει αυτή η απεριόριστη ποσότητα τέτοιων ε, τεμαχίων που φτάνει στην αγορά μας και που βέβαια είναι πολύ επιζήμιο κάτι τέτοιο για τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Αντιλαμβάνομαι ότι η γεωρική δομή είναι περίεργη στην Ουκρανία με τους ολιγάρχες και το ρόλο τους, ε, αλλά ε, για την Ουκρανία υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει Έχουμε και δύο στη Σλοβακία και Ολλανδία, διεθνή συνεργασία και από την Ευρώπη επωφελήθηκαν κάποιοι. Ε, δεν επωφελήθηκαν μόνο στην Ουκρανία. Ήταν ένα κόλπο, αλλά τέτοια κόλπα πρέπει να τα απομακρύνουμε, να μην επιτρέπουμε να υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε τη σαφή τη διάθεση να μην επιτρέψει τέτοιου είδου παραθυράκια. Θα δείχνει επομένω τη δέουσα προσοχή. Και όπω είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσπαθεί να αποκλεί τέτοιου είδου παραθυράκια και να προωθεί συμφωνίε που να μπορούν κάποιοι, να μην μπορούν μάλλον κάποιοι με κόλπα να καταχρώνται το σύστημα η, δι, η απάτη ε, θα υπήρχε. Ε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για απάτη εφόσον δεν είναι κάτι παράνομο, αλλά θέλουμε πιστή εφαρμογή της συμφωνίας. Και ελπίζουμε να μάθει το μαθημά της Ουκρανία. Και όπως είπε Πάμε και το επιβεβαιώνει η Κομισιόν να δωρεά γρήγορα από εδώ και πέρα για να αποφεύγονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Απαράδεκτες. Αυτό είναι και προς το συμφέρον των παραγών κρέατος πληρικών. Να μην φτάνουν τέτοιες απεριούσες ποσότητες ανεξέλεγκτες, γιατί αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός από πλευρά Ουκρανία. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω επίση να ευχαριστήσω του συναδέλφου ε, που συμφωνήσατε να μπει αυτό το θέμα στην μερίσια διάταξη ολομέλειας. Ελπίζω να μπορέσετε να κάνετε κάτι κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο δηλαδή της ε, Συνόδου Ολομέλειας του Νοεμβρίου να προσθεθεί αυτό το θέμα. Μια μικρή προσθήκη, έχετε μια ερώτηση, ναι. Κύριε Χάουταλα, δεν απάντησε ξεκάθαρα η Κομισιόν και εκπλήσωμε. Ούτε στην κυρία Γκρεγόρο, μεταξύ άλλων, απάντησε ξεκάθαρα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι δόλιο ή κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει απάτη ε, με αυτόν τον τρόπο κοπής και τι γίνεται με τις τελωνίκες αρχές των κρατών που έχουν εκδώσει νόμιες υποθέσεις ε, που επιτρέπουν αυτού του είδους ε, τη συναλλαγή. Στερικός έλεγχος από τη Γαμάλτα Σάνκο του Μαρτίου του 18. Ήδη εκεί αποκαλύπτονται παρατυπίες. Ελήφθη υπόψη αυτό ε, για να ληφθούν προληπτικά μέτρα. Λέτε δεν το περιμέναμε και μπάστα. Μα όχι, πρέπει να υπάρχουν προληπτικά μέτρα ε, και αποτρεπτικά μέτρα για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά μιλάμε και για την ίδια την αξιοπιστία της Ένωσης. Δεν ξέρω αν διαβάσετε τη Δευτέρα του New York Times. Διαβάστε τους. Κομισιόν, έχετε να σχολιάσετε κάτι, λέει ο Πρόεδρος. Ακούστε, για να κάνω μια ακόμη διευκρίνηση απάτη δεν υπήρχε σε σχέση με το πώς ενήργησαν οι τελωνιακές αρχές. Αυτό δεν ήταν παράνομο, ήταν σωστό. Εφάρμοσαν τις διαδικασίες που προβλέπονται. Δεν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό που έκαναν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και να επιμείνω για μια ακόμη φορά. Παρακολουθούμε, ελέγχουμε πολύ προσεκτικά την εφαρμογή της συμφωνίας. Έξω και σε πολύ πρώιμο στάδιο εντοπίσαμε το πρόβλημα και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να λαμβάνουμε μέτρα. Και έτσι ε, μπορέσαμε να το λύσουμε το πρόβλημα σε πρόωρο στάδιο. Σε πρόωρο στάδιο. Η Ναι, να απαντήσω και συγγνώμη που δεν αντέδρασα αυτό πριν. Σε καμία περίπτωση δεν θα κατηγορήσω ότι υπήρξε συνενοχή από πλευρά των Ευρωπαϊκών Τελωνιακών Αρχών όπως υπόθηκε, ήταν αυτό νόμιμο, γιατί έχουμε τους άλλους τρόπους τεμαχισμού. Τα άλλα τεμάχια μπορούσαν να φτάνουν ε, χωρίς καμία, ε, κανένα περιορισμό. Δεν φταίνε οι αρχές στα σύνορα για αυτά που έγιναν, γιατί ήταν νόμιμα. Απλά εκμεταλλεύτηκαν αυτό το παραθυράκι. Ήταν ένα κόλπο, ένα τέχνασμα που χρησιμοποίησαν. Δεν μπορούμε να το πούμε όμως απάτη. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν είναι ε, θεμητός ε, ανταγωνισμός αυτό που προέκυψε από την εφαρμογή αυτή της ε, συμφωνίας. Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι από τις κάτω χώρες, κύριε Σράιρ Πύρικ. Το 2018 και εγώ άρχισα να διαρωτώ ε, γιατί είπατε κι εσείς ότι εδώ δεν είναι αυτό που γίνεται απάτη. Το είπαμε στις κάτω και τώρα μας λένε ότι είναι νόμιμο αυτό από την Κομισιόν. Δεν έπρεπε να μας είχε ενημερώσει η Κομισιόν νωρίτερα. Κάναμε πολλή δουλειά και υπήρξε πραγματικά πολύ εκνευρισμός ε, στις κάτω χώρες. Πώς η Ουκρανία μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το νομικό κενό. Δεν μπορούσαμε να είχαμε ε, αντιδράσει πιο γρήγορα και να ήταν και πιο ξεκαθαρή απάντηση. Πράγματι πρέπει να αποφεύγονται τέτοια παραθυρά και είτε εννοούμε είτε παράνομα στι συμφωνίε μα, λέει ο πρόεδρο. Προθεσμία κατά των τροπολογιών τώρα. Λίγη σήμερα, στι 4 το μεσημέρι. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, μόνο στα αγγλικά παρακαλώ να καταθέσει τροπολογίε. Θα εγκρίνουμε στα τέλη του μήνα στη, την έκθεση στην Ολομέλεια. Θα ζητήσουμε να γίνει συζήτηση για τον Νοέμβριο. Όχι, έκανα λάθο λέει ο Θα ψηφίσουμε αύριο εμεί εδώ στην Επιτροπή μα και θα πάμε για την Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Άρα εδώ ολοκληρώνουμε το σημείο 4 και προχωρούμε με το... Συγγνώμη, το σημείο 5 και προχωρούμε στο σημείο 6, κατάσταση πρόοδου των ανεξέλιξης μέρων διαπραγματεύσεων, που δεν ε, είναι παρά μία αυτή η τριμερή διαπραγμάτευση που αφορά την αναδιατύπωση κανονισμού για τη διπλή χρήση. Ήδη από το 12 είναι ο κανονισμό. Τα τρία θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο, Κομισιόν, Συμβούλιο, συμφώνησαν να αναδιατυπωθεί ο λόγο κανονισμό, ώστε να ληφθεί υπόψη το γεγονό ότι υπάρχουν αυτέ τι τεχνολογίε πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για λόγους ε, κυβερνοεπιτήρησης και πρέπει να περιληφθούν στο κανονισμό διπλής ε, χρήση. Θέλουμε να ληφθεί υπόψη επίση η διάσταση τη ανθρώπινη ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα, έλεγχο εξαγωγών. Να έχει και αυτή τη διάσταση. Θέλουμε περισσότερο άνοιγμα, περισσότερη διαφάνεια μια πιο εναρμονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσέγγιση. Συμφώνησαν επ' αυτών των σημείων όλα τα θεσμικά και τα τρία. Χρειάστηκε πολύ καιρό όμως το Συμβούλιο να καταλήξει σε μια διαπραγματευτική εντολή. Ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς κάναμε τη δουλειά που είχαμε να κάνουμε. Και μετά από μακρές εντατικές συζητήσεις είχαμε στην ψηφοφορία 571 ψήφους υπέρ. Δεν ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και τώρα, μετά από πολλά χρόνια πλέον το Συμβούλιο, ξεκίνησε με την διαπραγματευτική εντολή και είχαμε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε και ο πρώτος τεμερής διάλογος έλαβε χώρα στις 20 Οκτωβρίου θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μα για να μα αναφέρει σχετικά ο κύριος Μπούχνερ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Όπω αναφέρθηκε, στην αρχή είχαμε μία μακρά καθυστέρηση, μέχρι δηλαδή να είναι πρόθυμο το Συμβούλιο να διαπραγματευτεί με εμά το πλαίσιο των τριμερών διαλόγων. Τώρα ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Οι θέσει όμως ε, είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Και όπως ήδη αναφέρθηκε, εμάς αυτό που μα απασχολεί είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, κατά την επιτήρηση, ε, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε ολοκληρώσει τις ε, πρώτες συζητήσεις που πήγανε πάρα πολύ καλά και ως εκ τούτου παρά τις διαφορές εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξο ότι δηλαδή θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Η Φινλανδική Προεδρία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα αυτό να ε, γίνει ταχύτατα και ενδιαφέρεται μάλιστα ενδεχομένως, ε, ενδεχομένως ε, να ολοκληρωθεί αυτό ο συμβιασμός κατά τη διάρκεια της δικής της Προεδρίας. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είμαι αισιόδοξο πρόεδρος. Περιμέναμε τέσσερα περίπου χρόνια για αυτή την εντολή για διαπραγματεύσει. και τώρα θέλουμε να τι ολοκληρώσουμε το των δυνατών. Ε, δεν ξέρω, μερικές φορές ε, πρέπει να είμαστε πιο ειλικρινεί και να εξετάζουμε ε, το θέμα επί της ουσίας. Πάντως, όπως πάντα, το πρώτο που παίζει ρόλο είναι η ασφάλεια. Ασφάλεια προηγείται της ταχύτητας, ε, όπως συμβαίνει και στις ε, μετακινήσεις. Ο επόμενος τριμμένος διάλογος προβλέπεται για τις 13 Νοεμβρίου. Κλείνει λοιπόν και το θέμα και πάμε στο θέμα υπαριθμών 7. Πρόκειται για, την, ε, για το ταξίδι στο Βιετνάμ που έλαβε χώρα η αντιπροσωπή αυτή μετέβη στο Βιετνάμ την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν αντιπροσωπή ad hoc και νομίζω ότι ήταν ε, μια πολύ επικοδομητική συνάντηση. Οκτώ πήγαμε, συμπεριλαμβανομένου του υποφαινόμενου. Είχαμε συναντήσει ψηλού επίπεδου στο Βιετνάμ. Μπορέσαμε να συναντηθούμε με όλους τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, ε, με κυβερνητικούς φορείς, με εκπροσώπους του Παγκόσμιου Γραφείου Εργασίας. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά. Πρώτα αποκτήσαμε μια εικόνα εκτός ε, κυβέρνησης και μετά ε, συναντηθήκαμε με τον Υπουργό ε, Βιομηχανίας και Εμπορίου, Υπουργό Εργασίας, ε, Υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων, με την Πρόεδρο της Βουλής, με μέλη της Βουλής Βουλευτές και τέλος συναντηθήκαμε και με τον Πρωθυπουργό. Και μπορέσαμε σε όλους αυτούς να θέσουμε τα θέματα που μας απασχολούν και που ε, συζητούνται σε σχέση με την εμπορική συμφωνία. Κατά την άποψή μου ήταν πολύ επικοδομητική αυτή η όλη επίσκεψη και για να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες θα δώσω το λόγο στον εισηγητή κύριο Σαραντήλ και βεβαίως είναι ευπρόσδεκτα και όλα τα άλλα μέλη της να προσθέσουν και εκείνα κάτι εφόσον το επιθυμούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας, ε, τη γραμματεία, το προσωπικό του συνεργάτες, Σταυμάσια η συνάντηση πολύ καλά οργανώθηκε και πήγε και πάρα πολύ καλά. Και μπορέσαμε λοιπόν να περάσουμε ένα πολύ καλό συμπυκνωμένο μήνυμα στους ε, Βιετναμέζους, ε, ε, σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Ε, νομίζω αυτό λήφθη υπόψη και όσον αφορά τα συμπεράσματά μας, ε, ειλικρινά σχεδόν σε όλες τις συναντήσεις ακούσαμε ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ είναι οι συμφωνίες αυτές απαραίτητες, ωφέλιμες, επωφελείς και πολύ χρήσιμες. Αυτό το είπε είπαν όλοι οι εκπρόσωποι της χώρας, ε, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το είπαν και εκπρόσωποι του Παγκοσμίου Γραφείου Εργασίας, το είπαν και ακτιβιστές με τους οποίους ε, συναντηθήκαμε, οι οποίοι είπαν ότι προσβλέπουν ε, στην επικύρωση της συμφωνίας, ότι οι στηρίζουν αυτή τη συμφωνία και τις αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν την ε, Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών. Ε, έτσι λοιπόν ε, η συμφωνία αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί θα ορίσει και συγκεκριμένε προδιαγραφές σε θέματα περιβάλλοντος. Επίσης θα βοηθήσει και στην διεθνή θέση του Βιετνάμ. Βεβαίω ακούσαμε ότι το Βιετνάμ θα μπορέσει να σημειώσει πρόοδο. Ε, το Βιετνάμ ε, θέλει να έχει καλή φήμη ότι τηρεί τις υποσχέσεις του και επίσης ε, θεωρώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το Βιετνάμ είναι μια επιτυχημένη ιστορία, είναι ένα success story. Έχει να παρουσιάσει εντυπωσιακά αποτελέσματα για την πρόοδο του τα τελευταία 30 χρόνια. Από την άλλη βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εξακολουθεί να είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα και δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα αυτά που επιθυμούμε εμείς να εφαρμόζονται χωρίς καθυστέρηση και στο ίδιο ακριβώς επίπεδο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τα συμπεράσματα, συμφωνώ με τον Πρόεδρο και με τους ε, συναδέλφους της αντιπροσωπείας ότι η εφαρμογή ο έλεγχος εφαρμογής της συμφωνίας ή και των δύο συμφωνιών που εγκρίθηκαν, αυτό είναι καθοριστική σημασία. Πρέπει να ελέγχουμε το τι ακριβώς εφαρμόζεται και το τι προβλέπει η συμφωνία και ίσως να ε, προσθέσουμε και νέα μέτρα εφόσον χρειαστεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω θα συζητήσουμε για όλα αυτά ε, με λεπτομέρειες ε, στην κοινή συζήτηση ευθύς αμέσως. Ε, παρακαλώ, μπορείτε κάλλιστα να μας πείτε τις απόψεις, να ακούσουμε και την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να ελέγχουμε προσεκτικά το ότι έγινε μετά την επικύρωση, να δούμε τελικά αν εγκρίθηκαν αυτά τα οποία επιθυμούμε και θέλουμε να επισημαίνουμε συνεχώς στους Βιετναμέζους ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά πόσο μπορούν να επιτύχουν περαιτέρω βελτίωση σε αυτόν τον τομέα. Αυτά είχα να σας πω προς το παρόν. Ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση. Ε, εκφράσαμε με απόλυτη ειλικρίνεια το τι περιμένουμε να γίνει, το τι επιτιμούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το τι θέλουμε να γίνει μετά την ολοκλήρωση της ε, επικύρωσης. Δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι οι Βιετναμέζοι δεν θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος, Μικλέ, ο κύριος Βίνκλερ και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και κύριε εισηγητή. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος, γιατί γρήγορα ε, ε, η σύντομη θα είναι η συζήτηση και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και εσάς Πρόεδρε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία στο, Χανόη, στο Ανόη και το διοικητικό προσωπικό που μας βοήθησε ιδιαιτέρως. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαμε ξαναπάει στο Ανόη και ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση. Στα Σπάργανα ήταν ο διάλογο μεταξύ Βιετνάμ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ μεγάλη είναι η πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Έχω την εντύπωση ότι πολλοί ουσιώδεις αλλαγές έχουν επέλθει στο Βιετνάμ καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ε, χρόνων που μεσολάβησαν μεταξύ των δύο επισκέψεων. Και θέλω να σας πω επίσης ότι κατά την άποψή μου η αλλαγή αυτή ε, ε, οφείλεται εν μέρη τουλάχιστον στο διάλογο που έχουμε κάνει με το Βιετνάμ και στις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και ναι, τη Συμφωνία Επενδύσεων. Πιστεύω ότι οι εταίροι που συναντήσαμε στο Βιετνάμ, στο Ανόη πιο συγκεκριμένα, γιατί, γιατί δεν πήγαμε και πουθενά αλλού, μόνο στο Ανόη μείναμε. Οι συναντήσεις λοιπόν με τους εταίρους μας ήταν πολύ καλές. Μια πολύ σημαντική συζήτηση έγινε με εκπροσώπους του, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ILO μας λέει ότι συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ανόη, στο Βιετνάμ και μας λέει ότι ουσιαστική πρόοδος έχει επιτευχθεί, έχει σημειωθεί και ότι επίσης φέτος κυρώνεται η μία από τις ε, τρεις ε, εκρεμείς συμβάσεις με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Έγινε αυτό και είναι πολύ σημαντική δέσμευση γιατί δείχνει δέσμευση στο υψηλότατο δυνατό πολιτικό επίπεδο και ο Υπουργό Εργασία του Βιετνάμ δεσμεύτηκε για το χρονοδιάγραμμα για την κύρωση των συμβάσεων ε, ε, και των δύο άλλων εκκρεμών συμβάσεων του χρόνου και το 2023 αντιστοίχω. Φέτο κυρώθηκε η πρώτη. Η Διεθνή Οργάνωση Εργασία μα είπε ξεκάθαρα ότι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και η κύρωση τη σύμβαση θα εκπληρώσει του στόχου τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία στο Βιετνάμ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είχαμε πολύ σημαντική συνάντηση με το Ευρωπαϊκό εμπορικό Επιμελητήριο στο Βιετνάμ, το οποίο μας παρασύωσε την κατάσταση πολύ ξεκάθαρα Πολλά μένει να γίνουν, πολλά εμπόδια έχουν αρθεί και θα μπορούσαν να είχαν αρθεί και χωρίς τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και χωρίς την Επενδυτική Συμφωνία, αλλά μένουν κάποια πράγματα πολύ σημαντικά που πρέπει να γίνουν. Αν δούμε τον ανταγωνισμό στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε ο μόνο σημαντικός παίκτη στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε, υπάρχει και η Κίνα, υπάρχει και η Ιαπωνία. Όμως, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Επιμελητηρίου, είμαστε οι μόνοι που έχουμε υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών στο Βιετνάμ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Κίρτον Ντάρλιν. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στη Γραμματεία και στην Αντιπροσωπεία. Ήταν εξαιρετική αποστολή, πολύ εξαιρετικά οργανωμένη. Το πρόγραμμα ήταν πολύ αποτελεσματικό, λειτουργήσε πολύ καλά. Την πρώτη μέρα ασχοληθήκαμε με τους μη κυβερνητικούς παράγοντες και αυτούς συναντήσαμε και ε, στο υπόλοιπο πρόγραμμα με τις επίσημες αρχές μπορέσαμε να στείλουμε ξεκάθαρα μηνύματα. Θέλω να συγχωρέω και εσάς κύριε Πρόεδρε για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάσατε τις ανησυχίες Αρχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μιλήσατε με ειλικρίνεια, σε κάποιες συναντήσεις μάλιστα με εξαιρετική ειλικρίνεια και καλά το κάνατε. Και ελπίζω πράγματι ότι ε, το πήραν το μήνυμα, σίγουρα το στείλαμε εμείς. Για να ολοκληρώσω την εικόνα, νομίζω ότι είναι δύο υπάρχουν δύο σημεία σημαντικά να πούμε. Το πρώτο, ναι, σε κάθε συνάντηση, είτε συναντιόμασταν με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, με μη κυβερνητικέ αρχές και συλλόγους και ενώσεις, με επίσημους ε, παράγοντες είχαμε την αίσθηση ότι η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και η Σύμβαση με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας θα βελτιώσουν το πλαίσιο των υφιστάμενων σχέσεων. Αυτό ναι, αλλά στις συναντήσεις με τις ΜΚΟ ακούσαμε ότι η κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ δύσκολη και μάλιστα επιδεινώνεται τα τελευταία χρόνια και αυτό πρέπει να το πούμε. Το ακούσαμε αυτό Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Είναι πολύ μεγάλες οι προσδοκίες από πλευράς οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στο Βιετνάμ. Πιστεύουν οι ΜΚΙ ότι αυτές οι συμβάσεις και συμφωνίες θα κομίσουν σημαντική αλλαγή και είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να την αναλάβουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να το εξετάσουμε προσεκτικά. Συμφωνώ με τον εισηγητή, με τον κύριο Ζαραντέλ ενδεχομένως να χρειαστεί να προβληματιστούμε ε, ποια έξτρα στήριξη μπορούμε να προσφέρουμε, πώς επιπλέον μπορούμε να στηρίξουμε αυτές τις συμβάσεις και συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ε, εξή θέμα που τέθηκε ήταν να φτιάξουμε ένα διακοινοβουλευτικό εποπτικό όργανο και αυτό το θέμα θα πρέπει να το πάρουμε ζεστά. Να δούμε πώς ε, το κεφάλαιο TST τίθεται σε ισχύ και επιβάλλεται υπό το φως της ε, θετικής ε, προόδου με το 98 υπάρχουν και ανησυχίες για τα εφαρμοστικά μέτρα. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί θα πρέπει να μπω στις λεπτομέρειες κάθε συμφωνίας. Όμως να τονίσω ότι η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, η ΜΚΟ, έχουν πάρα πολλές προσδοκίες από εμάς, άρα πολύ μεγάλη δική μας ευθύνη. Ναι, είναι υπέρ, αλλά είπαν ξεκάθαρα ότι η κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα επιδεινώνεται σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναλαμβάνω, και το χώρο που έχουν οι πολίτες να λειτουργούν. Ο κύριος Ντάντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για την πραγματικά εξαιρετική οργάνωση αυτής της ε, αντιπροσωπείας. Πάρα πολύ καλό το ταξίδι, σε πολύ υψηλό επίπεδο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι εγώ ήμουν πολύ επιφυλακτικός ε, όταν κάναμε τις προκαταρκτικές συναντήσεις. Ήμουν πολύ επιφυλακτικός για την κατάσταση που θα βρίσκαμε, αλλά γύρισα με δύο βασικά μηνύματα. Πρώτον, ότι όλοι με όσου όσους συναντηθήκαμε από την κυβέρνηση μέχρι και τις ε, οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών. Όλοι μας έδωσαν ένα σαφές μήνυμα ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε το Βιετνάμ σε αυτή τη φάση, πρέπει να τους στηρίξουμε γιατί καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, το είπε και ο συνάδελφος κύριος Βίνκλερ, ε, είδαμε τα στοιχεία που κατέθεσε και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, το να εγκαταλείψουμε το Βιετνάμ, αυτό είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το να το στηρίξουμε αυτή τη στιγμή. Προφανώς και υπάρχουν πολλά και σημαντικά θέματα τα οποία οφείλουμε να έχουμε κατά νου. Το άλλο μήνυμα που, θέλω, που πήραμε και θέλω να το μεταφέρω είναι να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τους διαλόγους. Δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα στις συναντήσεις ε, με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης ε, και με την κυβέρνηση και με τους εκπροσώπους ε, της κοινωνίας των πολιτών. Αυτά είναι τα θέματα που εξετάσαμε. Εγώ λοιπόν ε, έχω, έφερα μαζί μου και άλλη μια άποψη ότι υπάρχει μια πολιτική τάξη που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα ε, στο ποια είναι η άποψη της ε, κοινή ε, γνώμης. Το Βιετνάμ θέλει να προβάλλει μια καλή εικόνα στον κόσμο. Το Βιετνάμ θα ενταχθεί στο Συμβούλιο ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι αν θέλουν να παίξουν ένα διεθνή ρόλο, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη. Είναι δηλαδή σημαντικό να έχουμε μια συμφωνία με το Βιετνάμ. Προφανώς και εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα αλλά σε αυτή την νοτιοανατολική ε, περιοχή της Ασίας έχουμε το Βιετνάμ, ε, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει στο να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τους Κινέζους, αλλά και τα γεωπολιτικά θέματα της περιοχής που είναι πολύ σημαντικά. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά, λέει η κυρία Κάλσπρο, και να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέρτ Λάγκε, τον επικεφαλή τη αντιπροσωπεία μα, Να ευχαριστήσω τον Μάρτι Κάλρλο, την κυρία Κασκίνα, αλλά και την λυπή αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Βιετνάμ. Και όλου όσοι ε, είχαν καθήκοντα, του συναντήσαμε στο Ανόη και μας βοήθησαν. Ε, Χωρί αυτούς δεν θα είχαμε την ευκαιρία να μπορούμε να τα συζητούμε όλα αυτά τα θέματα. Ήταν συσκέψει και συναντήσει εξαιρετικά καλά προετοιμασμένε. Να σας πω ότι το εμπόριο με βάση τους κανόνες είναι κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη και την αηφόρο ανάπτυξη. Πράγματι ήταν πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα στο Ανόη, στο Βιετνάμ. Αποκομίσαμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση επιτόπου και είναι δύσκολο να μην εντυπωσιαστεί κανείς με την οικονομική πρόοδο και την ανάπτυξη του κλάδου της βιομηχανίας στο Βιετνάμ. Είναι πολύ αισιόδοξο το γεγονός ότι το Βιετνάμ θέλει να ενισχύσει το ρόλο του στη διεθνή κοινότητα. Μάθαμε ότι θα γίνουν βήματα για να κυρωθεί η Σύμβαση για τα Εργασιακά Δικαιώματα. Η πολιτική κατάσταση δυστυχώς δεν έχει αλλάξει και πολύ. Το Βιετνάμ παραμένει να συνεχίζει να μην είναι δημοκρατία και δεν μπορεί ο λαός να διαλέξει τον ηγέτη του. Δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ό,τι έχει να κάνει με την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του συνέρχεστε σε δημόσιο χώρο, αυτά δεν ισχύουν. Μπορεί να φυλακιστεί κάποιος χωρίς να έχει διαπράξει έγκλημα, αλλά να φυλακίζεται για τις σκέψεις του και υπάρχει και η θανατική ποινή στο ποινικό κώδικα και δεν έχει καταργηθεί η αντιπροσωπεία μας ήταν ξεκάθαρη ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι αποδεκτά. Τούτων λεχθέντων, ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ πρέπει να συνεχιστεί και οι συνάδελφοι του υπογράμμισαν άλλωστε οι διάφοροι εταιροί από την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, από τις ομάδες των ακτιβιστών με τους οποίους συναντηθήκαμε, πράγματι έχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουν να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο. Και αν εμείς πιστεύουμε ότι το εμπόριο είναι ένας δρόμος στην παγκόσμια αρένα για να που θα διασφαλίζει τη συνέχιση του διαλόγου, ε, τότε πρέπει να ε, το συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε αυτές τις ε, συζητήσεις. και να μην απογοητεύσουμε τους ακτιβιστές και ε, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρικμό είναι η επόμενη που έχει στο το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τον απολογισμό αυτή τη επίσκεψη που φαίνεται να ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Δυστυχώ δεν είχαμε τη δυνατότητα πράσινη να στείλουμε κάποιον. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε μια κοινή έκθεση των συμμετεχόντων που φαίνεται ότι ήταν πολύ καλή. Ε, είχατε ενδιαφέρουσες ε, συναντήσεις, αλλά νομίζω ότι οι εντυπώσεις μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με το συμμετέχοντα, άρα καλό θα ήταν να έχουμε ε, όλων τις απόψεις. Η ομάδα μας είχε ζητήσει να ακούσουμε εδώ κάποιον εκπρόσωπο από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και μας είπε ότι θα περιληφθεί αυτό στην ημερήσια διάταξη ε, όταν θα συζητήσουμε τον απολογισμό αυτής της επίσκεψης. Αλλά βλέπω ότι δεν συνέβη τελικά να έρθει ένας εκπρόσωπος από αυτή την οργάνωση. Θα ήταν νομίζω ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ροντρίγε Πινιέρο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση προς ε, τα μέλη της αντιπροσωπείας που ταξίδεψαν ε, στο Βιετνάμ και για την προηγούμενη που αναφέρθηκε ο κύριος Βίνκλερ. Η επιδείνωση που βλέπετε σε θέματα των δικαιωμάτων, ε, πώς την αισθανθήκατε, τι γίνεται με τις ΜΚΟ και τι σχέδια υπάρχουν ώστε γρήγορα να πάψει να ε, υφίσταται επιδείνωση της κατάστασης και των συνθήκων. Κύριο κύριος Λαντσίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Πραγματικά καταπληκτική ήταν η οργάνωση αυτής της αντιπροσωπείας και αυτού του ταξιδιού. Ε, πολύ καλά τα κατάφερε ο κύριος ε, Λάγκε ε, και επειδή έχω κάνει και άλλες αποστολές πραγματικά σας συγχαίρω. Λοιπόν, η Συμφωνία Ελεύθερων Ανταλλαγών με το Βιετνάμ και επειδή θα έχει και την Προεδρία στις χώρες Αζιάν είναι κάτι πολύ σημαντικό, ένα βήμα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την περιοχή. Κυρίως ε, έχοντας ε, κατά νου ε, τις επεκτατικές τάσεις της Κίνας και την αποτυχία της συμφωνίας με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θεωρώ ότι μπορεί πλέον να ανοίξει ένας χώρος για τις επιχειρήσεις και θέλω να υπογραμμίσω ότι όλοι όσους συναντήσαμε επί τόπου από τους πρεσβευτές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι και τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όλοι συμφωνούν ε, βεβαίως με αποχρώσεις ότι είναι απαραίτητο οι συμφωνίες να ολοκληρωθούν γιατί ε, προκύπτουν και οικονομικά και κοινωνικά Κα ωφέλη. Είναι βέβαια σαφές ε, ότι η άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα εργασίας και είναι σημαντικό αυτές οι συμφωνίες που θα συνάψουμε να βάζουν και κάποιες βασικές προϋποθέσεις που να μην είναι δυνατόν να γνωηθούν. Πρώτα απ' όλα θεωρώ το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό το θέμα ε, δεν μπορεί να αγνοείται. Ε, ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής μας, ο κύριος Λάγκε, ζήτησε να απελευθερωθούν 11 άνθρωποι που βρίσκονται στη φυλακή. Το ζητά αυτό ε, και η διεθνή κοινότητα. Ο κ. Λάμ, ο ε, Υπουργό Εσωτερικών, είπε ότι πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν παραβιάσει τον κείμενο ποινικό κώδικα, ο οποίο όμως ε, ποινικό κώδικα επιτρέπει και τη σύλληψη ανθρώπων απλά και μόνο γιατί εκφράζουν διαφορετική άποψη από αυτήν τη κυβέρνηση. κυβέρνηση. γίνονται βασανιστήρια, υπάρχει θανατική ποινή. Όλα αυτά βλέπουμε ότι ε, οδηγούν σε συμπέρασμα ότι υπάρχει καταστολή και καταπίεση. Η ε, κυβερνοεπιτήρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο για να ε, περιοριστεί η ελεύθερη έκφραση της άποψης, ελεύθερη έκφραση των πολιτικών απόψεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσει για όλα τα θέματα αυτά, γιατί είναι αξιολογήσει σε ε, τις οποίες θα πρέπει να κάνουμε με απόλυτη νυφαλιότητα, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα πούμε. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να υπάρχει και ε, προάσπιση των πνευματικών δικαιωμάτων, να προστατεύονται ε, τα εμπορικά σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από παραχάραξη. Το τρίτο θέμα που είναι σημαντικό είναι το περιβάλλον. Ε, στο Βιετνάμ η πρόεδρος ε, της ε, Βουλής, Εγγιουγέμ, δεν ξέρω τώρα αν το προφέρω και σωστά το όνομα, εν περιπτώσει αναφέρθηκε στο θέμα των παράνομων της λαθροθυρίας απλά και μόνο για ιδιωτικούς λόγους. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι επί το οποίο δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εμείς μέχρι τώρα έχουμε ακούσει μόνο καλές προθέσεις. Τώρα για την ε, ε, παράνομη υλοτομία και εκεί υπάρχουν ε, πάρα πολλές αντιρρήσεις, αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί από άλλες χώρες σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ο ποταμός Μανκόγκ έχει ρηπανθεί σε μεγάλο βαθμό, βεβαίως και με ευθύνη των Κινέζων. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει το πόσιμο νερό στο Βιετνάμ. Ε, το νερό αυτό σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιείται για τον ε, το ρύζι για να ποτίζουν τους οριζόνες. Μετά όμως ε, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα γιατί ε, δυστυχώς εξάγουν τις ποσότητες ρυζιού χωρίς όμως να υπάρχει ο έλεγχος και η τυποποίηση που προβλέπουν οι δικές μας οι που έχουν σχέση με τα βαρέα μέταλλα, τις χρωστικές ουσίες και ούτω καθεξής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ρήπανση του ποταμού Μανκόκ δεν σταματάει μόνο στα σύνορα του Βιετνάμ. Βλέπουμε ότι στους ωκεανούς υπάρχει υπάρχει το πρόβλημα των ε, πλαστικών στους ωκεανούς. Άρα δηλαδή τα πράγματα θα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους, ναι, να συνεχιστεί η συμφωνία, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και όλα αυτά τα θέματα που σας προανέφερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι έλεγχοι που γίνονται ε, θα πρέπει να γίνονται ακριβώς με τις ίδιες προγραφές όπως και σε άλλες χώρες και αυτό ας μην ξεχνάμε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει και σε σύγκρουση με την κυβέρνηση του Βιετνάμ. Άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν συστηματικοί έλεγχοι, ε, ταχεία εφαρμογή και όλα αυτά για να υπάρχουν εγγύησεις ότι γίνονται σεβαστές οι συμφωνίες, αλλά και για ε, να ε, είναι σαφής κατάσταση για όσους επιθυμούν στο μέλλον να συνάψουν συμφωνίες. Γιατί μην ξεχνάμε, όλα αυτά επηρεάζουν τη δική μας την ανταγωνιστικότητα, δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό ε, οδηγούν στο πρόβλημα της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς τώρα παρακαλώ, κύριε Χάταλ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσον ε, συστήσα το ζήτημα της εφαρμογής εθνικής νομοθεσίας που είναι και προϋπόθεση για να προωθηθεί η συμφωνία FLECT για τις ε, νόμες αγωγές ε, ξύλου. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που άπτεται τη συμφωνίας ελεύθερων ε, συναλλαγών, γιατί εκεί περιλαμβάνεται μνήα σε αυτή τη συμφωνία, στο κεφάλαιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείτε αυτή η εθελοντική συμφωνία εταιρική σχέσης για το ΦΛΕΚΤ. Η κατάσταση των δικαιωμάτων τώρα δεν βελτιώνεται, αντίθετα υπάρχουν σημάδια επιδείνωση. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό ε, έχει να κάνει με τον ποινικό κώδικο, όπως ακούσαμε τουλάχιστον. Πώς θέσατε το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων και τι απαντήσεις λάβατε στις παρατήρησεις σας. Είμαι βεβαία ότι θίξατε το θέμα αυτό, Πρόεδρος είναι να απαντήσω ίσως εκ της αντιπροσωπείας. Για το ΦΛΕΚΤ υπάρχει αυτή η δέσμευση, η επιβόλη δασικής νομοθεσίας διακυβέρνηση εμπορίου, αλλά και για τον νόμο περί κυβερνασφάλειας, Κάποιες υποθέσεις ε, για τον εντοπισμό, προστασία δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα και η πρόεδρος ε, της Εθνοσυνέλευσης είπε ότι θα πρέπει αυτή η εφαρμοστική πράξη να συζητηθεί με εμά, με το Ευρωκοινοβούλιο δηλαδή, ώστε να καταλήξουμε σε μια συνεννόηση μεταξύ μα. Υπήρξε λοιπόν δέσμευση ό,τι αφορά τη διαδικασία εφαρμογή για τα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα, πράγματι. Και εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ουσιαστική βελτίωση. Υπάρχουν άνθρωποι στη φυλακή επειδή έκαναν χρήση τη ελευθερία έκφραση αυτού του δικαιώματο. Αναμφίβολα. Όμως, και εκεί υπήρξε δέσμευση ότι θα εξεταστούν συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις. Και όπως λέτε και εσείς, φυσικά και το θέσαμε το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων. Νομίζω πως η συμφωνία μπορεί να φέρει και καλύτερες ε, δυνατότητες ε, συζήτησης κάποιων ζητημάτων στο πλαίσιο του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και φυσικά εμείς προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε ε, το μοχλό πίεση που μπορεί να έχουμε για να υπάρξει βελτίωση της κατάστασης στο Βιετνάμ. Είχα την δυνατότητα να περάσω το ΝΟΗ μια ακόμη μέρα συζητώντας ε, με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά αυτή την ε, συμβουλευτική ομάδα, την εγχώρια. όπου συζητούν ποιες είναι οι προσδοκίες τους, πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, την ομάδα αυτή τη συμβουλευτική και θα καταθέσουν αυτοί οι 25 φορείς ε, τις προτάσεις του σύντομα και εγώ είπα ότι θα τους υποστηρίξω στο διάλογο με την κυβέρνηση του Βιετνάμ. Να γίνονται σεβαστές αυτές οι ομάδες ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, γιατί το λέει και η συμφωνία. Εμείς τα τονίζαμε αυτά σε κάθε μας συνάντηση. Αυτές οι συμβουλευτικές ομάδες, 25 κτλ. Δεν πρέπει να θεωρούνται ως ε, ένας τρόπος συγκέντρωσης, ε, αλλά όλες οι ε, ομάδες κοινωνικών πρέπει να εκπροσωπούνται. Παραλαμβάνω λοιπόν ότι έγινε αυτή η συζήτηση και θα ξεκινήσει το παραπαρασκευαστικό έργο από την κυβέρνηση και είπαμε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, και οι συστάσει των συμβουλευτικών ομάδων των εθνικών για το περιβάλλον, για την εργασία. Και επειδή είπατε ότι υπάρχουν προσδοκίες, ναι φυσικά και υπάρχουν προσδοκίες. Ο κόσμος στο Βιετνάμ θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη συμφωνία για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης. Δήμεν. Ελπίζουμε να είναι θετικές λοιπόν οι πτώσεις της ε, συμφωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ που με επενέσατε για τον τρόπο με τον οποίο γύθηκα αυτή της αντιπροσωπείας. Επίσης να πω ότι όλοι σας ήταν στην ώρα σας, δεν καθυστερήσαμε σε καμία συνάντηση και γενικώ η επικοινωνία μας ήταν πάρα πολύ καλή. Είμαστε μια καλή ομάδα πιστεύω και να ευχαριστήσω ιδίω ε, το βάσμα, τη Βάσμα μάλλον που οργάνωσε αυτή την επίσκεψη. Ε, and, ε, yeah, this concludes, um, the... Και εδώ ολοκληρώνουμε το σημείο 7 και περνούμε ευθύ αμέσω στα σημείο 8 και 9 κοινή συζήτηση της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Ε, ε, σχέδιο σύστασης και σχέδιο έκθεσης. Αυτό είναι το σημείο 8 και 9. κύριος Ζαχράντη. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως εισηγητής χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι φτάσαμε επιτέλους σε αυτό το σημείο μετά από χρόνια διαπραγματεύσεων. Χαίρομαι και ελπίζω να έχουμε πράγματι φτάσει στο σημείο μη επιστροφής. Οι συνάδελφοι τόνισαν διάφορα ε, θέματα για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, Free Trade Agreement, είναι το πρώτο τέτοιου είδου κείμενο που εγκρίνει τον εκλεγέν κοινοβούλιο εδώ και αρκετό καιρό. Άρα και το τελευταίο, γιατί δεν έχουμε κάτι συγκρίσιμο το οποίο να ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Θα συμπληρώσει τις εμπορικές συμφωνίες που έχουμε ήδη συνάψει με άλλες χώρες της Ασίας. Θα θυμάστε τη Σιγκαπούρη, θα θυμάστε τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει το γεωπολιτικό ρόλο που της αναλογεί για άλλη μια φορά και να δώσει τον τόνο σε αυτό το ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον που απειλείται από τις εμπορικές εντάσεις. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρουσιάζεται ως πρωτοπόρο στην παγκόσμια εμπορική τάξη πραγμάτων δείχνουμε τη δέσμευση για ελεύθερο εμπόριο με βάση κανόνες, δίνουμε το σωστό παράδειγμα, δείχνουμε πόσα αυτά ε, επιφέρουν αμοιβαία ωφέλη, τα οποία δρέπουν οι κοινωνίες μας και πώς έχουμε ένα πολυμερές εμπορικό σύστημα με βάση τη μεταρρύθμιση του σχεδίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του ΠΟΕ. Αυτά καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, νομίζω ότι εδώ ε, διακυβεύεται η αξιοπιστία μας μπορούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι εταίροι, ότι διαπραγματευόμαστε αλλά και ολοκληρώνουμε και εφαρμόζουμε τις συμφωνίες μας και δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία να τα δείξουμε όλα αυτά. Να αναδείξουμε την αξιοπιστία, που έχουμε σε σύγκριση με άλλους παίκτες όπως είναι η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. γιατί αυτοί οι παίκτες δημιουργούν εμπορικές εντάσεις σήμερα ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τις κατευνάζει και αυτό είναι ένα παράδειγμα εξαιρετικό να προβάλλουμε παγκοσμίω στον υπόλοιπο κόσμο και πρέπει να υιοθετήσουμε αυτή τη ε, δέσμευση με τον Βιετνάμ και να τη στηρίξουμε απαρέγκλητα γιατί αλλιώ κάποιο άλλο θα έρθει να πάρει τη θέση μα. Νομίζω ότι ο κύριος Ντάντι και άλλοι συνάδελφοι το ανέφεραν αυτό, ότι οι παγκόσμιοι παίκτες ενδιαφέρονται ιδιαίτερως για τη χώρα αυτή και είναι έτοιμοι και καραδοκούν να έρθουν να καλύψουν οποιοδήποτε κοινό, κενό τυχόν αφήσουμε εμείς. Τρίτο πράγμα που θέλω να πω. Να αξιοποιήσουμε αυτή τη συμφωνία ως εργαλείο να προωθήσουμε τις αρχές μας. Η, Βιετναμέζη, η Βιετναμέζικη πλευρά θα πρέπει να κάνει αυτά που τις αναλογούν. Δεν πιστεύω ότι τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα θα βελτιωθούν εάν δεν εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία. Τι θέλει το ερώτημα αν δεν την εγκρίνουμε, τι θα έρθει να πάρει τη θέση της. Δεν νομίζω ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα. Και να θυμόμαστε ότι κατά βάση είναι μια εμπορική συμφωνία, όχι συμφωνία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί όμως να συμβάλλει ουσιαστικά και να επιφέρει αλλαγές στη χώρα. Ας μιλήσουμε ειλικρινά. Το ξέραμε, ακόμα και πριν αρχίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ξέραμε περί τίνο πρόκειται, τι συμβαίνει στο Βιετνάμ. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μέρος του συστήματος το οποίο αποκλίνει. Είναι πολύ μακριά από την ευρωπαϊκή δημοκρατία έτσι όπως εμείς την ε, ε, αντιλαμβανόμαστε. Και επιτρέψτε μου να σας κάνω μία προσωπική παρατήρηση. Είμαι 56 ετών. Τα πρώτα 26 χρόνια της ζωής μου τα πέρασα στην ε, κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα και το σύστημα εκεί ήταν πολύ παρεμφερές με το βιετναμέζικο σύστημα σήμερα. Πρέπει όμως να παραδεχτώ ότι το Βιετνάμ σήμερα είναι καλύτερο από αυτό που ήταν τότε η κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία. Ε, με, υπό πολλές πλευρές. Και πιστεύω πραγματικά ότι εάν τους δείξουμε το παράδειγμα και την καλή θέληση, καλή βούληση, τότε πράγματι θα έχουμε θετική απάντηση, ακόμα και στον τομέα και ιδιαίτερο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και τέλος, Συχνά λησμονούμε να τονίσουμε την οικονομική αξία αυτής της συμφωνίας. Είναι μια συμφωνία εμπορικών ανταλλαγών και πρέπει να αξιοποιήσουμε και να τονίσουμε τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα. Γι' αυτό και θέλω να τονίσω ότι αυτή η συμφωνία παρουσιάζει ευκαιρία, ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ανισορροπία σε ό,τι αφορά την εισαγωγή και την εξαγωγή αγαθών και αυτό πρέπει να αλλάξει. Η Βιετναμέζικη κοινωνία είναι δυναμική, έχει πολύ νεανικό πληθυσμό και πρέπει να περιμένουμε να τους εξάγουμε πράγματα. Είμαστε στην τέταρτη θέση, ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας, δηλαδή εισαγωγέας στο Βιετνάμ. Και δύο λόγια για το κείμενο για την διάλυση των εταιριών, Company Resolution. Χτίσαμε πάνω στη δουλειά που έχει γίνει στο παρελθόν. Ε, με έγγραφα που έχουν ήδη εγκριθεί και έχουν ήδη διατυπωθεί. Να τονίσω μόνο τα καινούργια στοιχεία. Με συγχωρείτε, διορθώνει η δερμηνέας, δεν είναι company resolution, είναι accompanying resolution, το ψήφισμα που συνοδεύει την έκθεση. Και ε, λέω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να ακυρωθούν δύο βασικές συμβάσεις, η 1.05 για την κατάργηση της εξαναγκαστικής εργασίας και η 87 για την ελευθερία του συνέρχεσθε. Το Βιετνάμ είναι σε πολύ καλή πορεία γιατί ακολουθεί την τροχιά της Σιγκαπούρης με, την οποία έχουμε ήδη κυρώσει εμπορικές συμφωνίες. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι η μεταρρύθμιση του εργασιακού κώδικα. Γίνονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό κώδικα. Το πιο σημαντικό έχει να κάνει με την εφαρμογή των συμβάσεων της, Διεθνής, ε, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Βλέπουμε εδώ έναν άμεσο αντίκτυπο που είναι αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Βιετνάμ. Συνεχίζεται αυτή η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την 21η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, με την οποία συναντηθήκαμε στο ΑΝΟΗ την περασμένη εβδομάδα και παραθέτω τα λόγια τους, το σχέδιο νέου εργασιακού κώδικα είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Συμφωνία Ελευθέρω Εμπορίου δίνει όθηση για τη δημιουργία μιας πραγματικά κοινωνικής και εργασιακής ατζέντα, δίνει την αίσθηση του επίγοντος και επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις. Τέλος της ποσό, ποσό της παράθεσης. Και σημαντικό είναι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τις σωστές ε, εργασιακές συνθήκες. Μπορώ να πω δύο λόγια για την εφαρμογή και υλοποίηση. Ο συζητητής Θέλω όλες οι συμφωνίες αυτές να προχωρήσουν και θα κάνω το παν προς αυτή την κατεύθυνση να έχω επικοδομητική συνεργασία. Περιμένω τις τροπολογίες σας, τις προτάσεις σας. Αυτά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thanks Σας ευχαριστώ. Τρία λεπτά ο κάθε σκιώδης εισηγητής. Ο κύριος Βίνκλερ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή, πολύ σοβαρός και αφοσιωμένος και το έργο του εξίσου καλό. Η οικονομική αξία της Συμφωνίας Έφερων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετναμ είναι προφανής. Πολλά νούμερα ακούστηκαν, αλλά πρέπει να δούμε και το γεωπολιτικό πλαίσιο. ΑΣΕΑΝ, καταρχάς, γιατί ρόλο θέλει να παίξει η σε αυτή την περιοχή. Και το Βιετνάμ σίγουρα ε, θα είναι σημαντικό εφαλτήριο. Και το δεύτερο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Δηλαδή, δεν μιλάμε για αμυγός εμπορικούς στόχους, αλλά για άλλα πράγματα τα οποία θα προωθηθούν χάρη στη συμφωνία αυτή εμέσως. Το πρώτο είναι οι συμβάσει ε, τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία και τα εργασία δικαιώματα εν γέννη. Ήθελα να το ελέγξω αυτό γιατί είχαμε μια συζήτηση ε, στο Υπουργείο ε, Εργασία στο Ανόη, όπου ακούσαμε ότι 15 εκατομμύρια εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή καλύπτονται από την εργασιακή νομοθεσία που ισχύει, αλλά μετά την τροποποίηση αυτού του νόμου θα επεκταθεί η κάλυψη. Θα τριπλασιαστεί ο ρυθμός των εργαζομένων που θα καλύπτονται με το νέο τροποποιημένο νόμο. Δηλαδή θα φτάσουμε στα 50 εκατομμύρια. Τεράστια πρόοδος. Επίσης μιλήσαμε για την κυβέρνο ασφάλεια. Είναι σημαντικό να υπάρχουν διατάξεις, νομοθεσία για την ε, ασφάλεια που να μην ε, αντιβαίνουν ε, με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις της Ένωσης στο βαθμό του δυνατού. Ελπίζω να το πετύχουμε αυτό. Επίσης, πολύ συζητήσαμε το φαρμαστικό σχέδιο, το πρόγραμμα εφαρμογής. Υπάρχουν προκλήσεις. Δεν υπάρχει κεφάλαιο για τις ΜΜΕ στη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Όμως πρέπει να προσέξουμε με τα διάφορα εργαλεία που πιστεύουμε θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρμογής και για την προστασία των ΜΜΕ. Αυτό λοιπόν το εργαλείο είναι μεταξύ άλλων ένα εργαλείο που θα οδηγήσει στην αλλαγή του Βιετνάμ. Οι μεταρρυθμιστές μπορούν να πάρουν νέες θέσεις. Έχουμε εκλογές το 2021 και δώστε μου 10 δευτερόλεπτα για να πω, όπως και ο εισηγητής, ότι και εγώ την ίδια ηλικία έχω με τον εισηγητή. Και εγώ τα πρώτα 25 χρόνια της ζωής μου τα έζησα σε μια σοσιαλιστική χώρα, λάθος, ε, στη λάθος πλευρά του σιδηρού παραπετάσματος. Άρα με άλλα μάτια βλέπουμε εμείς την πρόοδο στο Βιετνάμ. Και υπάρχει πραγματική πρόοδος, ναι, που όμως πρέπει να υποστηριχθεί από κάτι. Και αυτή η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών είναι ένας τέτοιος τρόπος για να στηρίξουμε το δυνάμει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αυτή είναι η δυνατότητα που έχουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν μεταρρυθμίσει στο Βιετνάμ μετά την ε, κύρωση. Το ξέρουμε από τι εμπορικέ συμφωνίε ότι η ισχύση του Ευρωκοινοβουλίου αλλάζει. Δηλαδή, ναι, μην μπορούμε να συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσει χωρί να έχουμε όμω τα χέρια μα στον ίδιο μοχλό Άρα, τους επόμενους μήνες πρέπει να τους ε, αξιοποιήσουμε με πολύ ε, προσεκτικό τρόπο και να είναι στρατηγικά τα αιτήματά μας. Πρέπει να φροντίσουμε οι ευρωπαϊκές αξίες να διέπουν ε, το διεθνές εμπόριο και να μην μένουμε στα λόγια αλλά και σε δράσεις, σε έργα. Αλλιώς δεν θα έχουμε την αξιοπιστία. Υπάρχουν προσδοκίες υψηλές από το λαό του Βιετνάμ Ακριβώ γιατί εμεί στέλνουμε το μήνυμα λέγοντα ότι η εμπορική μα πολιτική βασίζεται σε αξίε. Αν αυτό όμω δεν σημαίνει τίποτα, παραμένει στα λόγια, υπονομεύει τη δική μα την αξιοπιστία εν γέννη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί επαναλαμβάνω την προηγούμενη εβδομάδα στο Ανόη ακούσαμε διαρκώς και από αρκετούς σε διαφορετικές συναντήσεις που είχαμε ότι η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιδεινώνεται και είναι πολύ δύσκολο για τους πολίτες, ιδίως ό,τι αφορά την ελευθερία έκφρασης, ιδίως στο ίντερνετ. Αυτό μας το είπαν ξεκάθαρα. Νομίζω λοιπόν για αυτό το λόγο ότι η έκθεση του εισηγητού θα πρέπει να έχει ένα κεφάλαιο πιο έντονο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν νομίζω ότι περιλαμβάνονται αρκετά αυτή τη στιγμή στο κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση, πρέπει να επαναλάβουμε κάποια από τα αιτήματα που έχουμε διατυπώσει με πέντε ψηφίσματα ε, του Ευρωκοινοβουλίου από το 2013 μέχρι τώρα. 18 ε, δίκτυα ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων έχουν ε, δημοσιοποιήσει την αξιολόγησή τους για το Βιετνάμ και λένε ουσιαστικά τα ίδια πράγματα που λέμε και εμείς στα ψηφίσματά μας. Και τα ίδια ακριβώς αιτήματα πρέπει να τα επαναδιατυπώσουμε τώρα που είμαστε στη διαδικασία κύρωσης. Πριν εβδομάδα πάντως είδα ότι υπάρχει γνήσια διάθεση συμμετοχής και εμπλοκής των αρχών και τα λέγαμε αυτά ξεκάθαρα καταθέσαμε τα αιτήματά μας για την κυβερνοσφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα. Εκεί θα εστιάσω τις τροπολογίες μου. Εργασιακό δίκαιο και, ε, μετα... και τροποποίηση της εργασιακής νομοθεσίας. Αυτό στον νόμος πρέπει να τροποποιηθεί πριν ψηφίσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και εκεί πρέπει να περιλαμβάνονται οι διατάξεις των συμβάσεων 105 και 87 της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σε σχέση επίσης και με τον οδικό χάρτη. Πρέπει να έχουμε οδικό χάρτη για την αυτών των δύο συμβάσεων. Έχουμε 10 ε, εφαρμοστικά νομοθετήματα που επίσης πρέπει να εγκριθούν. Για το και δικαιώματα το είπα, είναι σαφής θέση του Κοινοβουλίου και πρέπει να την επαναλάβουμε και για τον νόμο περί κυβερνοασφάλειας. Ε, ο διάλογος συνεχίζεται και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ξεκάθαρα ποια θα είναι η εφαρμοστική νομοθεσία και τι αλλαγές ε, θα γίνουν προς την κατεύθυνση αυτής της νομοθεσίας για να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επανέρχομαι. Έχουμε μια σύντομη περίοδο στη διάθεσή μας, όπου μπορούμε να ασκήσουμε πίεση και πρέπει με πολύ στρατηγικό τρόπο να κινηθούμε πάνω σε αυτούς τους τρεις τομείς. Ήδη έχουμε θέσει στην επίσκεψή μας στο Βιετνάμ αυτές τις ανησυχίες. Έχουμε ε, ακούσει τι μας είπαν και καταγράψει τι μας είπαν και η ομάδα μας θα ψηφίσει ανάλογα με το τι θα έχει γίνει ώστε να δισκεδαστούν οι ανησυχίες μας στους τρεις αυτούς τομείς. Ευχαριστώ. Κάλσμπορ για την Renew. Το ερώτημα δεν είναι αν θα έχουμε ε, συναλλαγέ με το Βιετνάμ ή όχι, γιατί έχουμε ήδη συναλλαγέ σε μεγάλο βαθμό αυτή τη χώρα. Είμαστε ο τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο τη χώρα ήδη. Το ερώτημα είναι υπό ποιε προποθέσει, υπό ποιου όρου θα πρέπει να έχουμε συναλλαγέ. Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ε, βρήθη δυνατοτήτων και για τι δύο πλευρέ. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε για τον εμπόριο και τους κοινού για τι. Ε, δυνατότητε προ επιχειρήσει και Ευρωπαίου επιχειρηματίε για θέσει εργασία, για επενδύσει, καινοτομία, για τη βελτίωση των προτύπων, για τα εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον. Μπορούμε την εμπορική συμφωνία να την αξιοποιήσουμε με πάρα πολλού θετικού τρόπου, αρκεί να εφαρμοστεί σωστά αυτή. και αν υπάρχει διάθεση να υποστηριχθεί αυτή η συμφωνία και μετά την κύρωσή της. Και φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια Βιτναμέζους να έχουν πρόσβαση σε μία από τις πιο ανεπτυγμένες αγορές του κόσμου. Μιλούμε για μια χώρα που ήταν πάρα πολύ φτωχή για πολλά χρόνια, αλλά είναι ανοιχτή οικονομία, έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις οικονομικές και βλέπουμε πρόοδο στους ρυθμούς ανάπτυξης. Είναι πλέον μια χώρα που δεν πλήττεται πλέον από τη φτώχεια, αλλά το μήνυμά μας είναι σαφές. Έχουμε σαφείς ε, απαιτήσει ε, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα από τους Βιετναμίους φίλους μας. Και το έχουμε πει επανειμένως, το είπαμε και στο Ανόη, ότι είναι υψηλές προσδοκίες μας για αλλαγή στη χώρα. Και τώρα είναι η ευκαιρία τους και δική μας βέβαια, να συναντηθούμε σε ένα ισότιμο επίπεδο ως εταίροι. Και όλα αυτά τα λάβουμε υπόψη μας. Όταν ψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία στο Ευρωκοινοβούλιο. Η δημοκρατία όμως δεν γίνεται από μόνη της. Είναι δική μας ευθύνη. Πρέπει να κάνουμε εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε για να στηρίξουμε αυτή την εξέλιξη και η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών νομίζω ότι είναι ένας τρόπος. Αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός για να έχουμε στενότερη συνεργασία με το Βιετνάμ, θα δείξουν αυτή τη διάθεση άλλες χώρες. Αν πιστεύουμε ότι έχουμε ένα ρόλο να διαδραματίσουμε στο παγκόσμιο προσκήνιο, πρέπει να αναλάβουμε τι ευθύνε μα ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δείξουμε ότι αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε ευθυγραμμίζονται με τι αξίε μα. Ευχαριστώ. Uh, um, Ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρου των ε, Πρασίνων, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τη συνήθεια να έχουμε διαφορετικές ερμηνείες για την εφαρμογή και τον αντίκτυπο κάθε σε ελεύθερου εμπορίου και στην κατάσταση και ειδικά σε αυτό που μας αφορά σήμερα που είναι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμφωνώ με τη συνάδελφο κυρία Κίρτον Ντάρλιν. Τώρα έχουμε τους απαραίτητους μοχλούς για να ασκήσουμε πίεση και να προοδεύσει η κατάσταση στο Βιετνάμ. Το είπαμε και με ανακουφίζει που το ακούω, ότι δηλαδή παρόλο που ερμηνεύουμε διαφορετικά τα γεγονότα, συμφωνούμε όλοι στην εξή παραδοχή ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα η κατάσταση στη χώρα είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Το ίδιο εκφράστηκε και στην ακρόαση στην Επιτροπή ΔΟΑ νομικών υποθέσεων. Στην αρχή των διαπραγματεύσεων και υπόθηκε άλλωστε αυτό, ε, ε, τέθηκε το θέμα των πολιτικών κρατουμένων. Αυξήθηκαν κατά 50% οι πολιτικοί κρατούμενοι από την έναρξη των διαπραγματεύσεων μέχρι τον περασμένο Ιούλιο. Πριν από ένα χρόνο το Κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα ζητώντας την απελευθέρωση των συγκεκριμένων πολιτικών κρατουμένων. Και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης μας έχει επανειλημμένως ενημερώσει για το γεγονός ότι ο χώρος για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών συρρυκνούνται. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εκφράζει την ανησυχία της για τον περιορισμό της ελευθερίας του τύπου και διαδικτυακά και εκτός διαδικτύου ε, για ε, το ότι δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για την άμεση απελευθέρωση όλων των blogger ε, και όλων των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα μήνα πριν την υπογραφή. Και η κατάσταση δεν έχει εξελιχθεί. Δεν έχει προοδεύσει, δεν έχει βελτιωθεί. Δεν βλέπω να υπάρχουν αυτά στην έκθεσή σας, κύριε Ζαχραντήλ, και λυπούμε γι' αυτό. Νομίζω ότι έχετε δουλειά να κάνετε και θα πρέπει να τροποποιήσετε το κείμενο που μας έχετε υποβάλει, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από τα θέματα εμπορίου και των επενδύσεων. Το 2016 με μεγάλη πλειοψηφία, κατά δύο τρίτα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δοτήσει μια έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπινών δικαιωμάτων και στη δημοκρατία στον υπόλοιπο κόσμο. Και πάλι εκεί απευθύνουμε έκκληση για την θετική και συστηματική εισαγωγή ρητρών και διατάξεων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλε τι εμπορικέ συμφωνίε και επενδυτικέ συμφωνίε. Καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μηχανισμό απριόρι ελέγχου πριν από τη σύναψη κάθε συμφωνία ελέγχου δηλαδή για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να αποτελεί αυτό απαραίτητο και αναπόδραστο στοιχείο κάθε εμπορική σύμβαση. Εκλεγήκαμε πριν από έξι μήνε και λιγότερο. Είναι το, η πρώτη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου που, που εγκρίνουμε και συμφωνώ μαζί σα. Να μην είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο των φιλοδοξιών μα. Κρίμα είναι. Να δώσουμε νέα πνοή στι εργασίε μα. Και γι' αυτό θέλω να υποβάλω το αίτημα να μετατεθεί χρονικά η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ε, είναι πολύ σύντομες οι προθεσμίες αυτές. Υπάρχει και το Domestic Advisory Group, το χώριο συμβουλευτικό όργανο. 11 ε, Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, δεν φτάνει ο χρόνος. Με ενδιαφέρει η έκθεση αυτή, οι απαντήσεις για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε το ότι ο εργασιακός κώδικα στα μέσα Νοεμβρίου ε, θα υπάρξουν αλλαγές. Θα έχουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς νέα για την παιδική εργασία στο Βιετνάμ. Όλα αυτά θα πρέπει να τα έχετε για να μπορούμε να δουλέψουμε με σοβαρότητα και να τροποποιήσουμε το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαντσίνη παρακαλώ. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα θα πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και του περιβάλλοντος. Γιατί αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Δεν μπορούμε να τα κουκλώσουμε για γεωπολιτικούς και οικονομικούς ε, λόγους. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η κατάσταση και πρέπει να έχουμε τη σιγουριά ότι θα υπάρξει βελτίωση. Ακόμα και αν είναι μια χώρα που τηρεί τις υποσχέσεις της, ε, πρέπει να έχουμε τη σιγουριά ότι αυτές οι υποσχέσεις ε, θα τηρηθούν, ε, θα εφαρμοστούν αυτά που υποσχέθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος, γιατί αυτή είναι η δική μας η πολιτική, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ερμηνεύει τον κόσμο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η τροπολογίες ε, μπορούν να βοηθήσουν το Βιετνάμ έτσι ώστε να ακολουθήσει την πορεία που επιθυμούμε όλοι μαζί από κοινού. Σας επαναλαμβάνω ότι η συμφωνία είναι σημαντική, αλλά ε, όλα αυτά ε, θα πρέπει να επιμείνουμε στο να προβληθούν οι δικές μας οι και αυτές ε, να επικρατήσουν οποιονδήποτε οικονομικών συμφερόντων από πλευράς κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Μορέλ για την ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συγητής είπε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Βιετνάμ έχουν διαρκέσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και αληθές είναι αυτό, αλλά εμείς ως κοινοβουλευτικοί έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να διαβάσουμε ένα κείμενο, να το τροποποιήσουμε και να το ψηφίσουμε. Συμφωνώ με την εκπρόσωπο των Πρασίνων να μετατεθεί χρονικά για αργότερα η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, γιατί πολλά αγνοούμε και πολλά δεν μας έχουν ανακοινωθεί σήμερα, μέχρι σήμερα. Όντω, η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου δεν είναι μόνο οικονομική. Υπάρχει μια αμυγό πολιτική διάσταση και εγώ προσυπογράφω πλήρω το στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση των Πολιτικών να ενισχύσει τι σχέσει τη με το Βιετνάμ και τι λοιπέ χώρε σε αυτή την περιοχή, την τόσο σημαντική από γεωπολιτική σκοπιά, δεν το αφισβητώ. Όμω, Υπάρχει και η οικονομική σκοπιά. Κατάλαβα τα συμφέροντα τη αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία ικανοποιείται ιδιαίτερω με τη συμφωνία. Κατάλαβα τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών που πιστεύουν ότι θα έχουν πρόσβαση στου διεθνεί και δημόσιου διαγωνισμού στη χώρα αυτή. Αλλά δεν θα είναι τόσο εύκολο με την προθεσμία των 15 ετών. Έστω όμω, καταλαβαίνω ότι θέλουν να πάρουν μεγάλα δημόσια έργα. Όμως, ποιο είναι το συμφέρον του Ευρωπαίου καταναλωτή, του Ευρωπαίου εργαζόμενου, του Βιετναμέζου εργαζόμενου, του Βιετναμέζου πολίτη. Δεν ξέρω γιατί αυτή η συμφωνία τους ωφελεί. Και το βλέπω αυτό και στα ψηφίσματα και στην άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι χαίρονται γιατί είναι το Βιετνάμ μια πλατφόρμα συναρμολόγησης για τις χώρες της Ασίας. Ακόμα και οι Κινέζοι χρησιμοποιούν τους Βιετναμέζους για τα νέα εργαστήρια αλλά δεν θα πρέπει εμείς να χαιρόμαστε γιατί ο κίνδυνος είναι η μετεγκατάσταση, ακόμα μεγαλύτερη και περισσότερη μετεγκατάσταση στον τομέα της μεταποίησης και δεν νομίζω ότι αυτό είναι καλό για τον Ευρωπαίο εργαζόμενο. Τώρα, για τον καταναλωτή, ας μην είμαστε υποκριτές. Ε, το κεφάλαιο για την ε, αηφόρο ανάπτυξη είναι πολύ ελαφρύ. Απουσιάζουν οι κανόνες και ποιότητα, η χνηλασιμότητα των προϊόντων. Μιλήσαμε για λαθρέα, για παράνομη αλληλεία. Ε, διάφορα προβλήματα δεν έχουν ρυθμιστεί. Είναι η χώρα που μολύνει τα με πλαστικά τον ωκεανό και είναι στη τέταρτη θέση του μεγαλύτερου ρηπαντή στον κόσμο. Έχουμε και το Λάος και την Καμπότζη που ε, στέλνουν ξυλία παράνομη πολύτιμη στο Βιετνάμ και ε, συμβάλλουν στην αποδάσωση και αποψήλωση των δασών. Και μετά λέμε να σεβαστεί η Συμφωνία των Παρισίων, όπου ε, και εκεί δεν είναι σωστή η διατύπωση. Άρα για τη διατροφική επιστημιστική ασφάλεια, για τον κίνδυνο υπερεκμετάλλευση, για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Εκεί υστερούμε πάρα πολύ και υστερούμε πάρα πολύ και για τους εργαζομένους, Ευρωπαίους και Βιετναμέζους. Χαίρομαι κύριε εισήγητη, γιατί είσαστε ειλικρινέστατος και είπατε ότι δεν είναι συμφωνία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ, το καταλάβαμε. Αλλά δεν είπαμε ότι είναι συμφωνία ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θα νύψουμε έτσι τα σχήρα μα και θα πούμε ότι δεν μα νοιάζει. Και το είπαν και οι προηγούμενε ομιλήτρε. Η κατάσταση το μόνο που κάνει επιδεινώνεται. Ε, θα, κάνουμε, θα κλείσουμε τα μάτια, θα κάνουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Μιλούμε για παιδική εργασία για συνθήκες εργασίας αυτή τη στιγμή στο Βιετνάμ, ε, ε, τα οποία ε, δεν έχει υπογροθεύσει καθόλου η κατάσταση, το αντίθετο κιόλας. Δεν συμμερίζομαι τον ενθουσιασμό σας και ζητώ να έχουμε περισσότερο χρόνο να εργαστούμε, να τροποποιήσουμε και να έχουμε πιο απτές και συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Έχουμε λοιπόν άλλους 7 που έχουν Ζητήστε λόγο η κυρία Πεγκίνη Τιτσιάνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Κοιτάξτε, όσον αφορά την εμπορική πολιτική, είναι απόλυτα σαφές ε, ότι οι στόχοι είναι κυρίως οικονομικοί. Όμως αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα εργαλείο για να προάγουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο. Και βεβαίως μόνο εφόσον το αποφασίσουμε αυτό. Υπάρχουν και τα θέματα τα οικονομικά, γιατί ε, Τελικά ε, είναι αλήθεια ότι το Βιετνάμ προσφέρει τεράστιες ε, ευκαιρίες στους δικούς μας επιχειρηματίες, 4 εκατομμύρια άνθρωποι, πολύ μεγάλο ποσοστό ανάπτυξης. Από την άλλη βέβαια είναι σαφές ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα, από, σε όλο αυτό το διάστημα που δεν εφαρμόζονταν οι δικοί μας οι κανόνες, αυτό ε, δημιουργεί πρόβλημα ανταγωνιστικότητας στις επιχειρήσεις μας. Άρα δηλαδή αυτή η συμφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από προπολογισμό προϋποθέσεις. Ε, μία εξ αυτών προφανώς και είναι η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή μου κυρίως στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, στην περίπτωση αυτή δεν ξέρω, δεν κατάλαβα καλά. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης αναστολή εφαρμογής της ε, συμφωνίας και δεν ξέρω αν το κατάλαβα καλά, ίσως μπορείτε να μου απαντήσετε. Ε, άλλο θέμα, το θέμα του οι δικές μας οι επιχειρήσεις έχουν ήδη υποφέρει από εισαγωγέ ε, ρυζιού από την Καμπότζη και το Βιετνάμ. Ίσως θα πρέπει να υπάρχουν και εκεί ε, κάποιες ε, δικλείδες ασφαλείας. Ε, τελειώντας, θα ήθελα να πω ότι κατά τη δική μου τη είναι απολύτως απαραίτητο ε, να τεθεί αυτή η συμφωνία σε εφαρμογή, αλλά με δύο προϋποθέσεις. Ε, πρώτον, η μία προϋπόθεση αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεύτερη αφορά την προστασία της γεωργίας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να, κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή και τους ειδησκιώδεις και όλους όσοι συνεργάστηκαν για αυτή τη δουλειά, η οποία είναι σημαντική για να υπερασπιστούμε τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να βοηθήσουμε το Βιετνάμ σε αυτή τη μετάβαση ε, σε μια σύγχρονη οικονομία με αηφόρο ανάπτυξη που θα έχει αναλάβει αυτή τη δέσμευση και θα έχει αναλάβει και τη δέσμευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, Αξιολογώ και κρίνω θετικά την πρόοδο από τις, ε, που έχουν σημειώσει οι Βιετναμέζικες αρχές. Ξέρετε, είχατε 25 χρόνια εμπειρία, λέτε, με το σιδηρούν παραπέτασμα στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία και εμείς είχαμε 40 χρόνια τη δικτατορία του Φράγκο και ξέρουμε τι σημαίνει η καταστολή της ελευθερίας του λόγου και τι σημαίνει να είσαι πολιτικός κρατούμενος. Νομίζω ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως στις ε, δημοκρατικές αρχές, την ελευθερία της έκφρασης και γι' αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν θα γίνουν τα απαραίτητα βήματα για να υπάρξει αυτή η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με οποιοδήποτε εμπορικό μας εταίρο. Θα δώσουμε ε, προτιμησιακή πρόσβαση. Με ανησυχούν διάφορα θέματα, όμως πώς θα καταφέρουμε να γίνει η σωστή αξιολόγηση με πλήρη εκπροσώπηση της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στις εθνικές συμβουλευτικές ομάδες. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ελεύθερα συνδικάτα και σωματεία, πώς θα εγγυηθούμε για την ε, αντιπροσωπευτικότητα όλων των συνομιλητών μας, ότι εκφράζουν αντιπροσωπευτικά την κοινωνία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η κυρία Βαν Μπρέμπτ. Ε, και εγώ να επανέλθω στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, προφανώς ε, το θέμα των συμφωνιών ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών το θέμα είναι ότι όλοι θα θέλαμε να έχουμε με χώρε που έχουν τα δικά μα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά το άλλο θέμα που είναι πιο σημαντικό είναι τι θα κάνουμε με χώρε όπου επιδεινώνεται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντί να βελτιώνεται. Εμεί ε, έχουμε μία τέτοια συμφωνία ε, με το Βιετνάμ από το 2014. Έκτοτε όμω η κατάσταση αντί να βελτιωθεί έχει επιδεινωθεί. Γι' αυτό έχω μία ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί υπάρχει μία σχέση ανάμεσα στο PCA και το FTA, τη Συμφωνία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στο Βιετνάμ, να το πω έτσι πολύ απαλά, δεν και ιδιαίτερα καλή. Γι' αυτό ερωτώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκεί που γίνεται λόγο στην παράγραφο για την συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, τι ακριβώ σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιο θεωρεί ω κριτήριο για να χρησιμοποιήσει τη ρήτρα που προβλέπει τη σύνδεση αυτών των ε, θεμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να αξιολογήσουμε την Συμφωνία Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών που μας έχει κατατεθεί. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ εκείνους ε, που πήγαν με την αντιπροσωπεία ε, στο Βιετνάμ. Εγώ πήγα εκεί πριν από κάποια χρόνια ε, κάποιοι λένε ότι κατ' ουσίαν πρόκειται για ζούγκλα, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Δουλεύουν πολύ σκληρά, βλέπουν τα πράγματα κάτω από διαφορετική οπτική γωνία και ε, νομίζω ότι ε, θα πρέπει να δούμε κάπως διαφορετικά το θέμα της ε, Συμφωνίας ε, Ελεύθερων Εμπορικών Ανταλλαγών. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πολλή δουλειά και από τις δύο πλευρές, και από την Επιτροπή και από την πλευρά του Βιετνάμ, κυρίως όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχουν βέβαια επιφυλάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτό το κατανοούμε. Δεν πρέπει να επιδεινωθεί η κατάσταση, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Βίνκλερ, ω εισηγητής και οι δύο συγητές κατ' ουσίων επισημαίνουν ότι η χώρα δεσμεύτηκε ότι θα επιχειρήσει κάποια βελτίωση. Όπως αναφέρθηκε, η γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή αυτή και το παγκόσμιο εμπόριο ε, περιλαμβάνει και τη Σιγκαπούρη βέβαια που και αυτή είναι πύλη προς τις υπόλοιπες ε, χώρες της ε, ΑΖΕΑΝ. Το να έχουμε εμπορικές ανταλλαγές με τη Σιγκαπούρη και να απορρίπτουμε με το Βιετνάμ, αυτό δεν έχει νόημα ούτε πολιτικά ούτε από οποιαδήποτε άλλη σκοπιά. Έχουμε λοιπόν μια πολύ σημαντική συμφωνία. Η αντιπροσωπεία που πήγε εκεί ε, πρέπει να μας πει τι ακριβώς έμαθε, τι πληροφορήθηκε αν απολύπταμε τη συμφωνία, πρέπει να διορτηθούμε αυτό σε τι θα βοηθούσε και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Η κυρία Χάουταλα. Ε, κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι κατ' ουσίαν δεν διαφωνούμε για το τι ε, θα θέλαμε να κάνει το Βιετνάμ πριν ή μετά την επικύρωση αυτής της συμφωνίας. Εκεί που μοιάζει να διαφωνούμε είναι το ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να ασκήσουμε πίεση. Και συμφωνώ με κάποιον που είπε προηγουμένως ότι δεν είναι τώρα ε, κατάλληλη η χρονική στιγμή. Δεν πρέπει να τα περάσουμε πολύ γρήγορα όλα αυτά από το Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχουν κάποια ε, θετικά δείγματα από πλευράς Βιετνάμ ότι θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση. Γιατί λοιπόν ε, δεν δίνουμε στο Βιετνάμ την ευκαιρία να προχωρήσει. Θα ήθελα λοιπόν να στηρίξω αυτό που ελέγχθη προηγουμένως, ότι θα πρέπει να τους δώσουμε λίγο χρόνο, μέχρι την επόμενη χρονιά, αρχές της επόμενης χρονιάς. Υπάρχει η υποεπιτροπή αυτοποιών δικαιωμάτων, που και αυτή προετοιμάζει μία γνωμοδότηση, εκεί είμαι σκιώδη συγγήτρια και νομίζω ότι από αυτήν την υποεπιτροπή θα προκύψουν ε, χρήσιμες ε, προτάσεις ε, για το τι είδου μηχανισμοί είναι απαραίτητοι για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Βίνκλερ, αυτό το παράδειγμα που αναφέρετε δεν είναι απόλυτα πιστικό. Γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το παράθυρο για μεταρρυθμίσεις στη Ρουμανία ήταν ανοιχτό μέχρι να γίνει η Ρουμανία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν εξελίξεις που δεν είναι απόλυτα ικανοποιητικέ. Ε, για το Βιετνάμ ε, το παράθυρο είναι το ανοιχτό, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή και την πόρτα. Κύριος Μπορλά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, να τον συγχαρώ για τη σκληρή δουλειά που έκανε για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Εμείς θα στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία ανεπιφύλακτα για τρεις λόγους. Πρώτον, είναι εμπορική η συμφωνία. Ο εισηγητής το υπογράμμισε αυτό. Ε, θα ενισχυθούν οι εξαγωγές μας και θα ενισχυθούν και οι εξαγωγές του Βιετνάμ. Το 2035 προβλέπεται ότι θα έχουμε αύξηση κατά 19% των εξαγωγών μας, 8 δις ευρώ ε, αύξηση της ανάπτυξης για τους Βιετναμέζους, 15 δις ευρώ. Αυτά είναι τα στοιχεία, αυτά ε, θέλουμε να επιτύχουμε εάν ε, καταργηθούν όλοι οι δασμοί και πολλά άλλα εμπορικά εμπόρια, εμπόδια θα έρθουν και αυτά. Άρα δηλαδή η ε, νέα ε, δυναμική κοινωνία του Βιετνάμ θα στηριχθεί, ε, θα έχει μεγαλύτερη βημερία και κοινωνική πρόοδο. Δεύτερον, αναφέρθηκε ότι από γεωστρατηγικής πλευράς είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να είναι παγκόσμιος παίκτη να είναι παρούσα στην περιοχή. Ε, η απάντηση στον προστατευτισμό είναι το ελεύθερο εμπόριο και αυτό ρυθμίζεται με τις ελεύθερες εμπορικές ανταλλαγές. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, η βιωσιμότητα, νομίζω αυτό είναι ένα καθοριστικό στοιχείο της συμφωνίας. Είναι τα πράγματα τέλεια? Προφανώς και δεν είναι τέλεια. Υπάρχει πρόοδος που πρέπει να την επιβλέπουμε. Αυτό είναι πρόεδρο, θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ ε, θεωρώ ότι πρέπει να συσταθεί μια διακοινοβουλευτική επιτροπή. Ε, κύριε Πρόεδρε. Θέλω όμως να σας ερωτήσω μήπως υπάρχουν τροπολογίες και από άλλες επιτροπές, ας πούμε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κύριος Ντάμπτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω δύο θέματα. Πρώτον, όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το Βιετνάμ ε, είναι μια χώρα όπου παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου τα δικαιώματα εργασίας είναι ιδιαίτερα επισφαλή, έτσι να το πω και εξοραίζοντας την κατάσταση. Εγώ νομίζω το ε, πιο σημαντικό είναι ότι ξέρετε ποιοι είναι οι πιο επιφυλακτικοί ε, σε αυτή τη συμφωνία, τα συνδικάτα. Ε, η πολιτική είναι πολύ πιο ανοιχτή, αλλά τα συνδικάτα αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικά. Θέλω να πω το εξής. Είναι πολύ δύσκολο να ε, προσπαθούμε μέσα από μια εμπορική συμφωνία να προσπαθούμε να αλλάξουμε ε, το Βιετνάμ και να το κάνουμε δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή στο Βιετνάμ έχουμε μονοκομματική κυβέρνηση, μονοκομματική πολιτική κατάσταση. Ε, παρόλα αυτά πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα τα εργαλεία που μας προσφέρει η εμπορική πολιτική και αυτή η συμφωνία έτσι ώστε να γίνουν σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Και τα εργαλεία που έχουμε έχουμε στα χέρια μας σε αυτή τη φάση. Αυτά τα εργαλεία πρέπει ε, να ξεκαθαρίσουμε, να προβάλλουμε ποια είναι τα αιτήματά μας. Τι το καλό θα προκύψει από αυτή τη συμφωνία, από τη στιγμή που θα ε, εγκριθεί. Ε, τι περιμένουμε, ε, τα πολιτικά δικαιώματα, τα συνδικαλιστικά, τα εργασιακά δικαιώματα και την κυβερνοασφάλεια. Γιατί και η κυβερνοασφάλεια έχει άμεση σχέση με τις δικές μας τις επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια στο Βιετνάμ. Κατόπιν υπάρχουν τα θέματα των πολιτικών ε, το πώς εφαρμόζονται ορισμένα πράγματα. Ε, essential clause. Αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο, αυτή τη ρήτρα ε, γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο κατά τη φάση της εφαρμογής της συμφωνίας μας προσφέρει τις εγγύσεις που περιμένουμε από το Βιετνάμ. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή ο κύριος Βάρμπορν συνολικά, το λέω αυτής εξ αρχής, τη στηρίζω τη συμφωνία. Με πιο συλλογιστικό, με πιο σκεπτικό. φοβούμαι μην μείνει πίσω η Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα. Είναι σοβαρό το θέμα και το παρατηρούμε να συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες. Αν δούμε πριν 10 χρόνια, τετραπλασιάστηκε η οικονομία της Κίνας 81% αύξηση και στο Βιετνάμ, ε, Ινδία περίπου στα ίδια, ενώ η Ευρώπη 16-17%. Άρα μένουμε πίσω δυστυχώς και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μεγάλη ευημερία μακροπρόθεσμα, θα έχουμε πιο μικρή ανταγωνιστικότητα ε, για τις επιχειρήσεις μας. Δεν αυξάνεται όμως μόνο η Ασία, αυξάνονται και οι ΙΠΑ με ταχύς ρυθμούς, ταχύς ε, σχεδόν όσο το Βιετνάμ. Άρα χρειαζόμαστε αυτή τη συμφωνία προκειμένου να μπορέσουμε εμείς να ευημερίσουμε. Γιατί πρέπει οι εταιρείε μας να μπορούν να πουλούν τα προϊόντα τους στην αυξανόμενη μεσαία τάξη του Βιετνάμ. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία και πρέπει να τη στηρίξουμε το συντομότερο δυνατόν. Διότι κάθε μέρα χάνουμε σαν ανταγωνιστικότητα. Άρα είναι πήγον να κυρωθεί η συμφωνία. Λείπει κάτι όμως από αυτή τη συμφωνία. Ένα κεφάλαιο της ΜΜΕ. Ελπίζω στη φάση της εφαρμογής να μπορέσουμε να εργαστούμε από αυτού, ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας να μπορούν να εξάγουν και να εισάγουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ο Κρίστοφ Χάνσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και εγώ ε, τον εισηγητή για την ε, πάρα πολύ καλή του δουλειά. Πράγματι πρόκειται για μια στρατηγική για εμάς συμφωνία για την ε, χώρα αυτή της περιοχής ΑΣΕΑΝ. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός και θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπουρζουά ότι πρόκειται για εμπορική συμφωνία. Δεν είναι ένα ε, καλά στο οποίο μπορούμε να βάλουμε τα πάντα και να λύσουμε όλα τα προβλήματα του κόσμου όσοι πήγαν στο Βιετνάμ είδαν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτελεστεί στο πλαίσιο της ΔΟΕ, της Σύμβασης 98 ε, που έχει κυρωθεί και επίσης έχει αναγγελθεί και τροποποίηση του εργασιακού νόμου. Επομένως όλα αυτά ε, δείχνουν άλματα πρόοδου και σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε ό,τι αφορά το περιβάλλον για παρα... και εκεί η χώρα προσπογράφει τη συμφωνία στον Παρισινό για το κλιματικό θέμα δηλαδή. Άρα τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο κύριος Μορέλ είπε πρόκειται μόνο για μια συμφωνία που θα ωφελήσει την βιομηχανία. Δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Μορέλ. Υπάρχει και ο αγροδιατροφικός τομέας που υποφελείται πάνω από 160 γεωγραφικές ενδείξεις προστατευόμενες αναγνωρίζονται πλέον με αυτή τη συμφωνία και χθε το βράδυ είχαμε μια εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο ακριβώς ε, ε, του Σπαρμεζάνα, σες Γκοργκοντζόλα, του Κοντέ, του παραγωγή αυτών των, τυριών ε, περιμένουν από εμάς να τους προστατεύσουμε από παραποιημένα προϊόντα και την, το σφετερισμό της ε, διανοητικής τους ιδιοκτησίας. Είναι μια αναψώμενη χώρα, το Βιετνάμ θα τους βοηθήσουμε, θα τους δώσουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία με την συμφωνία αυτή για να κάνουν σημαντική πρόοδο, αυτό δεν το ξεχνάμε. Είμαι υπέρ της ε, αναβολής, ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη υποθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. Ευχαριστώ. Και στρέφομαι τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ελένα Κένια, την αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ Εμπόριο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και Ζαχράντιλ. Με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα τα αποτελέσματα της, ε, τον απολογισμό της αποστολής στο Βιετνάμ. Ήταν ανοιχτό, είπατε και ειλικρινή, ο διάλογος, με χαροποιεί αυτό. Και εμείς το ίδιο διαπιστώνουμε όταν έχουμε συναντήσει υψηλό επίπεδο με τους Βιετναμέζους, ότι υπάρχει μια ειλικρίνη και ένα άνοιγμα στις επαφέ μας. Θα ήθελα να εστιάσω σε διάφορους τομείς στην παρέμβασή μου, αρχίζοντας από τις οικονομικές πτυχές που αναφέρατε αρκετοί και είναι σίγουρα και η βάση οποιασδήποτε συμφωνίας ε, ελευθέρων συναλλαγών. Είναι μια φιλόδοξη συμφωνία στο ίδιο επίπεδο με αυτήν που έχουμε με τη Σιγκαπούρη που είναι ήδη μια πολύ πιο ανοιχτή αγορά από ότι το Βιετνάμ. Πέραν των δασμών καταργούνται όλοι οι φραγμοί ένθεν κακήθεν. Υπάρχει κάποια διαφορά σε ό,τι αφορά την περίοδο εφαρμογής, γιατί είναι, όπως είπα, αναπτυσσόμενη χώρα το Βιετνάμ, αλλά μετά το πέρας ε, της δεκαετίας ε, θα έχουμε πλήρη κατάρριξη των δασμών. Όπως γνωρίζουμε βέβαια, οι οικονομικές πτυχές ε, του εμπορίου αφορούν πολύ περισσότερο τα πρότυπα, την εύκολη πρόσβαση στις αγορές, την προστασία της, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Όλα αυτά καλύπτονται από αυτή τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών στο ίδιο υψηλό επίπεδο ε, όπως και με χώρες όπως η Σιγκαπούρη. Η προκειμένη συμφωνία όμως δεν, ε, το παραλαμβάνω θα οδηγήσει ε, σε μια δυνατότητα να περνάνε τα κινέζικα προϊόντα στις ευρωπαϊκές αγορές. Δεν ενδιαφέρονται να είναι ε, μια χώρα διαμετακόμισης για την Κίνα, το Βιετνάμ, ξέρουν ε, γιατί έχουν επαφές με, το, με τη χώρα αυτή ε, και σίγουρα δεν θα θέλουν να μπαίνουν τα κινέζικα αγαθά στη χώρα τους και μέσω αυτής στις δικές μας. Αλλά και εμείς θα το δούμε και θα δούμε και τις κινέζικες επενδύσεις και πώς προχωρά αυτό το θέμα. Ένα άλλο θετικό με αυτή τη συμφωνία είναι ότι δεν υπάρχουν ε, ε, σημαντικές γεωργικές σε εμπορικέ μα συναλλαγέ με το Βιετνάμ για τον Ιταλό βουλευτή. Ναι, το ρύζι είναι ένα ευαίσθητο θέμα με το Βιετνάμ, όμως έχει ξεκαθαριστεί η ποσότητα ε, του ρυζιού που μπορεί να μπαίνει αδασμολόγητα στην Ένωση. 30.000 τόνοι ρυζιού. Επίσης, σε τα πρότυπα, έχουμε δεσμεύσεις σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα. Οπότε μπορούμε εύκολα να εξαγάγουμε αγαθά ε, στο Βιετνάμ. Αυτό θα ωφελήσει όχι όμως μόνο τις μεγαλύτερες, αλλά και τις μικρές, τις ΜΜΕ, που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σίγουρα στα διάφορα πρότυπα που ισχύουν στις ε, κάστοτε χώρε. Για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ένα σχόλιο συγκεκριμένα. Πράγματι διαπραγματευτήκαμε τη συμφωνία αυτή πριν ε, θεσπιστεί αρχή να υπάρχει σε όλες τις συμφωνίες ελευθέρων των αλλαγών κεφάλαιο τη ΜΜΕ. Όχι ότι δεν υπάρχουν όμως διατάξεις για τις ΜΜΕ. χάρη, διαφάνεια, πρότυπα για την είσοδο τα κτλ. Όλα αυτά περιλαμβάνονται. Αλλά όταν περάσουμε στην φάση της εφαρμογής, θα το δούμε πολύ ξεκάθαρα. Και θα δούμε τι εργαλεία έχουν στη θέση μας, ώστε οι ΜΜΕ και από τις δύο πλευρές να επωφεληθούν πλήρως της συμφωνίας. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα των αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναφέρθηκε από πολλούς. Ξεκινώ από το σκέλος των αξιών. Έχουμε το κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και περιλαμβάνεται τα περί αξιών εκεί, όπως και με όλες τις συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε. Έχουμε τέτοια διατάξεις και υπάρχει δέσμευση για την ε, συγκρότηση των ε, εθνικών συμβουλευτικών ομάδων για χώρε όπω το Βιετνάμ. Ναι, αυτό θα αποτελέσει πρόκληση. Όμως, όπως ε, ορισμένοι από όσοι πήγαν στην επίσκεψη αυτή στο Βιετνάμ διαπίστωσαν και το κομμουνιστικό κόμμα θα πρέπει να ακούει αυτές τις ενώσεις, αλλά υπάρχουν και άλλοι από την κοινότητα των πολιτών που ενδιαφέρονται και είπαμε ξεκάθαρα στις αρχές του Βιετναμού ότι περιμένουν να είναι ανοιχτέ αυτές οι συμβουλευτικές ομάδες ώστε να περιλαμβάνουν συνολικά την κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν κάποια ζητήματα ε, που είναι πιο λεπτά σε ό,τι αφορά το Βιετνάμ. Που έχουμε κάνει το, το κόμμα και την επιβιωσή του, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ΜΚΟ περιβαλλοντικές ή δραστηριοποιούμενε σε άλλους τομείς που θα θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτές τις εγχωρίες ε, συμβουλευτικές ομάδες. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο υποστηρίζει αυτές τις ομάδες. Εμείς ήδη συνεργαζόμαστε με το Βιετνάμ για να συμβεί αυτό. Για την παιδική εργασία, ένα σύντομο σχόλιο είναι σίγουρα μια προτεραιότητα και της νέας Κομισιόν και της νέας ε, Προέδρου της Κομισιόν. Η παιδική εργασία έχει επισημανθεί ως μείζον πρόβλημα στο Βιετνάμ. Υπάρχει μια έρευνα για την επικαιροποίηση των στοιχείων που είχαμε πριν από πέντε χρόνια και από τη ΔΟΕ επίσης, Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, ε, ε, έχουμε στοιχεία που λένε ότι έχει μειωθεί ε, δραματικά η εργασία κατά 50%. Τέλο πάντων θα έχουμε κάποια στοιχεία το Δεκέμβριο μάλλον. Και υπάρχει και δέσμευση εκ μέρους του Βιετνάμ ότι θα καταρτήσουν ένα πρόγραμμα εργασίας για την εκρίζωση τη παιδική εργασίας και θα συνεργαστούν μαζί μας στο μέτωπο αυτό. Ένα σημαντικό σημείο, εμείς στηρίζουμε, έχουμε το πρόγραμμα υποστήριξη προς το Βιετνάμ, και θα συνεχίσουμε να το έχουμε για την ε, εφαρμογή της συμφωνίας δεν αφορά μόνο τη χρήση των μηχανισμών που έχουμε, αλλά και την υπαρχή υποστήριξη για τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να περιλαμβάνει σε όλες τις συμφωνίες. Ναι, πράγματι. Όμως αυτή τη συμφωνία έχουμε άμεση ε, σύνδεση με τη Συμφωνία Τερξίας και συνεργασία. Δεν ισχύει με όλες τις χώρες, αλλά με το Βιετνάμ ισχύει ότι υπάρχει αυτή η άμεση διασύνδεση και μπορούμε να αναστείλουμε τη συμφωνία. Ακριβώς λόγω της ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν υπάρχει ε, κάποιο σημείο αναφορά, ε, benchmark, γιατί δεν ξέρουμε πού να το βάλουμε σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι θέμα από το που προέρχεται κανεί, ε, αλλά αν υπάρξουν δείγματα σοβαρή επιδείνωση, αυτό θα είναι ένα θέμα συζήτησης και είμαι βέβαια ότι και το Κοινοβούλιο θα δώσει τη προσοχή. Και ολοκληρώνοντα να πω το εξή. Αυτή η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών είναι ένα ακόμα λιθαράκι στο σύνολο αυτών των μηχανισμών που έχουμε και συμφωνιών με το Βιετνάμ για να μπορέσει το Βιετνάμ να προχωρήσει αυτό που εμεί θεωρούμε ότι είναι σωστή κατεύθυνση, δηλαδή άνοιγμα, ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα και έρχεται να προσθεθεί στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας. Έχουμε και την ε, διαδικασία Αγιουγιού για την παράνομη λαθρέα αναρχιαλία, τη Συμφωνία Φλέγκτ και βέβαια παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά από πλευράς Κομισιόν την εφαρμογή. Ευχαριστώ. Κύριε Ζαχράντιλ, θέλετε κάτι να προσθέσετε. Uh, thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, ίσως ε, να πω κάποια λόγια στο θέμα που αφορά στην εφαρμογή της ε, συμφωνίας και Ίσως υπάρχουν κάποια πράγματα που να ξέχασα στην αρχική μου παρέμβαση. Το ψήφισμα υπογραμμίζει την καθοριστική σημασία της εφαρμογής, την εφαρμογή της συμφωνίας και τονίζει το ρόλο ε, του ειδικού ε, συμβούλου αυτού που θα ασχολείται με θέματα εμπορικά. Υπογραμμίζει ε, επίσης και το ρόλο του νέου επιτρόπου σχετικά με την παροχή τεχνικής αρρωγής. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι καθοριστική σημασία να ελέγχουμε την εφαρμογή της συμφωνίας από τις αρχές του Βιετνάμ, κυρίως όταν πρόκειται για την εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί φοβάμαι ότι αυτό σίγουρα θα είναι πρόβλημα. Κατά τα άλλα, να πω και κάτι άλλο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δεν κάνω λάθος, ε, έχουμε και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, η οποία γνωμοδότηση αυτή θα μπορούσε ε, να συμπεριληφθεί στο ψήφισμά μας και νομίζω ότι ε, το θέμα ε, καλύπτεται ικανοποιητικά, καλύπτονται όλες οι πτυχές ε, της ε, παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Τέλος, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η συμφωνία υπογράφηκε πριν από τέσσερα χρόνια. Κατ' ουσίαν ήταν το Δεκέμβρη του 2015. Έκτοτε λοιπόν το κείμενο δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Η μόνη αλλαγή που έγινε αφορά στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και εκεί αναφέρεται ότι το θέμα των επενδύσεων πρέπει να αφαιρεθεί από τη συμφωνία, να εξεταστεί ξεχωριστά, γιατί ε, υπάρχει μεν κάποια αρμοδιότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η ουσία της συμφωνίας παραμένει ίδια. Αυτό ήθελα να πω. Και επίσης να πω ότι λόγω ε, επιβαρημένης ημερήσιας διάταξης ε, της Ρουμανικής Προεδρίας κατά το πρώτο εξάμεινο αυτού του έτους ε, δεν μπορέσαμε να εξετάσουμε το θέμα της συμφωνίας. Δεν μπορούσαμε να την εξετάσουμε τη συμφωνία πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε εγκρίνει αυτή τη συμφωνία πριν από τις εκλογές, δυστυχώς αυτό έγινε μετά, έγινε τον Ιούνιο, τότε θα είχαμε ήδη να κάνουμε μία ε, συμφωνία ε, που θα μπορούσε να συζητηθεί ε, κατά διάρκεια των, της προεκλογικής Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι υπέρ του να αναβάλουμε πράγματα. Ε, πιστεύω ο συγητής ότι θα πρέπει να τηρήσουμε το αρχικό χρονοδιάγραμμα και δεν βλέπω ε, το τι θα μπορούσε να προκύψει κάποιο όφελος από ε, περαιτέρω αναβολή. Τέλος, ως εισηγητής θέλω να σας αναφέρω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερα για να επιτευχθεί ο στόχος και να δουλέψουμε μέσα σε ένα φιλικό και επικοδομητικό πνεύμα, να συνεργαστώ με όλους σας όταν θα ε, κατατεθούν ενδεχομένω τροπολογίες ή κάποιες επιθυμίες σας για αλλαγές σε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα της εφαρμογής της συμφωνίας προφανώς και είναι καθοριστική σημασίας. Εγώ είπα να συσταθεί μια επιτροπή ελέγχου ε, που θα παρτίζεται ε, και από πλευράς Βιετνάμ, από την Πρόεδρο της Βουλής, από εκπροσώπους του Βιετνάμ και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μια τέτοια επιτροπή ε, για να εξετάζει το όλο θέμα και από κοινοβουλευτική σκοπιά. Υπάρχει τώρα διορία 11 Νοεμβρίου, 5 ώρα το απόγευμα, είναι καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. Μετά ε, θα περιμένουμε τις γνωμοδοτήσεις από τις επιτροπές που θα γνωμοδοτήσουν Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, Επιτροπή Ανάπτυξης, Συντέβε και η Επιτροπή Ελίας. Και μετά θα έχουμε περαιτέρω συζητήσεις για το ψήφισμα, για τις ε, τροπολογίες, για τις ε, γνωμοδοτήσεις των επιτροπών. Αυτά θα γίνουν στις 2 και 3 Δεκεμβρίου και φαντάζομαι σε αυτές τις ε, συναντήσεις ε, θα προσκαλέσουμε εκπροσώπους ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και εκπροσώπους από το Βιετνάμ. Κατόπιν θα ακολουθήσει η περίοδος των Χριστουγέννων, θα τα σκεφτούμε και πάλι και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου έτσι ώστε το όλο θέμα να πάει στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Και πάμε τώρα στο δεύτερο τμήμα στο θέμα των επενδύσεων. Ο κύριος Ζαραντήλ. Θα είμαι πολύ σύντομος κύριε Πρόεδρε. Ε, γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά γιατί έχουμε να εξετάσουμε αυτό το κομμάτι της συμφωνίας το οποίο αρχικά ήταν ενταγμένο μέσα στην συμφωνία κανονικά, στο σύνολο της συμφωνίας, αλλά λόγω απόφασης που λήφθη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγκαστήκαμε να το αφαιρέσουμε. Βεβαίως αυτό που ενδιαφέρει είναι η ίση όρη ανταγωνισμού, αλλά ας είμαστε ειλικρινεί, κάποια πλευρά θα είναι σε καλύτερη θέση για να επενδύσει στην άλλη πλευρά. Και προφανώς αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ αυτή η συμφωνία προσφέρει τεράστιες δυνατότητες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως στον τομέα των δημόσιων διαγωνισμών. Ε, η οικονομία του Βιετνάμ αναπτύσσεται ταχύτητα με ρυθμό ανάπτυξης 5,1%. Ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια για να γίνουν επενδύσεις στην υποδομή. Ακούσαμε από την κυβέρνηση του Βιετνάμ ότι επιθυμεί να αυξήσει την συνεργασία της ε, με τον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις. Έτσι λοιπόν αυτή η συμφωνία που προτείνεται ε, θα διευκολύνει τις επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Βιετνάμ. Ε, πρόκειται λοιπόν ε, για ε, προσθήκη στην συμφωνία. Εγώ θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα στηρίζω και θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και πάλι να συνεργαστώ με όλους εσάς για να ολοκληρώσουμε αυτό το συγκεκριμένο ψήφισμα. Προσβλέπω λοιπόν στα σχολιά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό λοιπόν τους σκιώδους εισηγητές να είναι όσο σύντομοι όσο και ο εισηγητής, ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. 21 χώρες μέλη έχουν διμερείς επενδυτικές συμφωνίες με το Βιετνάμ, οι οποίες θα καταργηθούν όταν η νέα συνολική επενδυτική συμφωνία τεθεί σε ισχύ. Πιστεύω ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι όσο δεν το πιο ανοιχτό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει η Επιτροπή να το προσέξει πολύ αυτό το ζήτημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίσης, θέλω να στηρίξω την πρότασή σας, κύριε Πρόεδρε, την οποία υποβάλατε στο Βιετνάμ και επαναλάβατε εδώ στην Επιτροπή μας. Η τρέχουσα ομάδα παρακολούθησης με τον ένα με τον άλλο τρόπο μπορεί να συγχωνευτεί ή, εν πάση να μεταμορφωθεί σε ένα εποπτικό όργανο εμείς ως ΕΛΚ στηρίζουμε αυτή την ιδέα, είναι μια πολύ καλή ιδέα και στηρίζουμε και την επενδυτική συμφωνία με το Βιετνάμ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Τζούντ Κίρτον Ντάρλιν. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω τα σχόλια που έκανα για τη συζήτηση για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, αλλά βεβαίω συνεχίζουν να ισχύουν και συνδέονται και με την επενδυτική συμφωνία, με το IPA και με το FTA. Οι επενδυτικές ροές ήταν πολύ με σημαντικές για την οικονομική ανάπτυξη του Βιετνάμ. Το μάθαμε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης την περασμένη εβδομάδα και οι επενδυτές επενδύουν περιμένοντας ότι δεν θα τους πάρει κανείς ε, την περιουσία χωρίς αποζημίωση. Έχουμε κάποιε μελέτε από την UNTAD για την προστασία των επενδυτών και έχουμε και το σχέδιο έκθεση του εισηγητή το οποίο λέει ότι το ICS θα ενθαρρύνει τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και την επενδύσει με αυτόματο τρόπο. όμω εγώ νομίζω ότι πρόκειται για ευσεβεί πόθου. Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ ISTS και επενδυτικέ ροέ, Ρώτησα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μου απάντησαν γιατί βάσει στοιχείων δεν υπάρχει σχέση ε, αιτίο, αιτία του μεταξύ των δύο. Υπάρχουν 82 που δεν έχουν ISTS με το Βιετνάμ παρά τις σημαντικές ροές FTA ε, ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Και παρόλο που οι επενδυτές θέλουν το ISTS ή το ICS, δεν το χρειάζονται κατά κύριο λόγο. Άρα το θεμελιώδες ερώτημα που ζήτεται είναι η δικαιοσύνη σε σχέση με την καταστρατήγηση του νόμου, η δίκαιη αντιμετώπιση. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν πρέπει να την χάνουν διακρίσεων σε σύγκριση με τις βιετναμέζικες επιχειρήσεις. Έτσι όμως δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το νόημα. Το ICS κάνει διακρίσεις υπέρ των διεθνών συνεργασιών και δημιουργεί ένα ξεχωριστό νομικό σύστημα για αυτές, ενώ τα συμφέροντα των περιβαλλοντολόγων, των εργαζομένων, των ακτιβιστών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαρτώνται από τη δικαιική τάξη και την ένομη τάξη εντός της χώρας του Βιετνάμ. Και παρόλο που ε, μπορεί να υπάρχουν καταστρατηγήσεις, αυτές δεν θα τύχουν των ακυρώσεων που θα τύχουν οποιαδήποτε παραβίαση γίνει σε σχέση με τα δικαιώματα των διεθνών στρατηγικών επενδυτών. Είναι πολύ μικρή η ισορροπία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωμη Τάξη θα πρέπει να εμπλέξουμε τις πολυεθνικές, να πιέσουν, να επιφέρουν αλλαγές στην εσωτερική δικαστική τάξη στο Βιετνάμ, έτσι ώστε να ωφεληθούν και οι εγχώροι ακτιβιστές και υπέρμαχοι ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ επόμενη ομιλήτρια για το Ρινιού. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξαιρετικές της επιδόσεις και τη Σεσίλια Μάλστρομ και τον επικεφαλής διαπραγματευτή. Η κύρωση αυτής της συμφωνίας δεν είναι ένα θέμα του κατά πόσο θα πρέπει να επενδύσουμε ή όχι στο Βιετνάμ. Ήδη οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύουν πολύ, χωρίς τις εγγυήσει που να τους προσφέρει μια διεθνής επενδυτική συμφωνία. Αν υπάρξει όμως θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις επενδύσεις τους και να τις αυξήσουν, να τις αναπτύξουν με ένα σαφές πλέγμα κανόνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει αυτή την επικοινωνία. Ο, το εμπόριο, οι επενδυτικές συμφωνίες είναι πολύ σημαντική συνιστόσα για ανοιχτές κοινωνίες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τούτων λεχθέντων. Να πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και να μην υποτιμούμε το νόμο μας ως νομοθέτη και όχι ως υπαγόμενο σε κανόνες στην παγκόσμια οικονομία. Εμείς βάζουμε τις τους κανόνες, δεν υποκύπτουμε σε αυτούς και αν δεν το κάνουμε εμείς και θα έρθει κάποιο άλλος να πάρει τη θέση μας. Πρέπει να έχουμε ισχυρές θέσεις για τις προσδοκίες μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ. Πρέπει να τρέφουμε υψηλές προσδοκίες έτσι ώστε να γίνουν τα βήματα για τη βελτίωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα δεν βοηθά. Uh, Ευχαριστώ. Η κυρία Πρίκμο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η συμφωνία εδώ αναφέρεται στα κεφάλαια για την αεφόρα ανάπτυξη και στην οικονομική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν αλλάζει και τίποτα. Άκουσα ε, προηγουμένως ότι όλοι θέλουν να δουλέψουν με την έννοια της δέουσας επιμέλειας, due diligence. Και ο Επίτροπος Χόγκαν έχει μιλήσει γι' αυτό. Άρα η συμφωνία μπορεί να επεκταθεί, να πάει πολύ πιο πέρα από ό,τι προβλέπεται σε ό,τι έχει να κάνει με τους στόχους της αηφόρου ανάπτυξης. Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάινεν, η νέα πρόεδρος, επιμένει ιδιαίτερως για το θέμα αυτό. Άρα θα έπρεπε η συμφωνία να πάει παρά πέρα. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου το 2016, το Συμβούλιο επιμένει για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντό των επιχειρήσεων και να ληφθεί υπόψη αυτό ο, ο σεβασμό ε, σε, στην περίπτωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και έχουν κομμάτια τη αλυσίδα αξιών που εδράζονται και βρίσκονται στο εξωτερικό και υπάρχουν και νόμιμα μέσα προσφυγή και ό,τι έχει να κάνει με τι καταστρατηγήσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντό επιχειρήσεων. Άρα μπορεί να βελτιωθεί το κείμενο και η διατύπωσή του υπό αυτή την έννοια, γιατί πράγματα που υπάρχουν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου δεν υπάρχουν στη συμφωνία έχει υποθεί ξανά και ξανά ότι το Βιετνάμ είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα, τα συνδικάτα δεν είναι ανεξάρτητα, δεν έχουν ελευθερία λόγου, το δικαστικό σύστημα πόρο απέχει από το να είναι άρτιο, ο τοπικό πληθυσμό ή εργαζόμενοι πολύ δύσκολο μπορούν να λάβουν αποζημίωση οι εργαζόμενοι πολύ δύσκολα μπορούν να λάβουν αποζημίωση ή αποκατάσταση των προβλημάτων του και των παραβάσεων που τους, ε, από τι οποίε πλήττονται. Τώρα, μας έχει προβληθεί το εξής επιχείρημα. Ε, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος και δεν έχει γίνει αξιολόγηση. Ας δώσουμε χρόνο για να γίνει αυτή η αξιολόγηση. Είναι απαραίτητο ε, για θέματα δικαίου και δικαιωμάτων θεμελιωδών, για θέματα ένομης τάξης. Ως πράσινοι θέλουμε απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη των συμφωνιών, να υπάρχουν επαληθεύσιμα συμπεράσματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και για την κατάσταση για τη λαθρέα, την παράνομη αλία, την αποψήλωση των δασών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε 7 χρόνια διαπραγματεύσεις το να τη ζητούμε να δράσει σε λίγες εβδομάδες δεν είναι λογικό. Και επιτρέψτε μου, θα ακούσουμε τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο, αλλά τις ΜΚΟ δεν θα τις ακούσουμε εδώ σε ακρόαση. Δεν θα τους καλέσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ο κύριος Λαντσίνη, παρακαλώ στην ε, δική μου τη χώρα ε, πολλές φορές όταν δεν θέλει κανείς να ακούσει ε, λέει και ξαναλέει τα ίδια. Εγώ λοιπόν θέλω να ελπίζω ότι τελικά ε, πραγματικά θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά που είναι προβλήματα και τα οποία τα επισημάναμε από την αρχή. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένες πράξεις, συγκεκριμένα γεγονότα, αλλιώς θα συνεχίζουμε να μιλάμε, να λέμε διάφορα λόγια, αλλά δεν θα καταλήγουμε πουθενά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά θα τελεσφορήσουν. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, είμαι πολύ πειθαρχημένος, το γνωρίζετε. Δεν είναι νέο το ερώτημα, ούτε νέα η συζήτηση. Συμφωνώ με την Τζούντ. Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ επενδύσεων και αυτά που μας υπόσχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή τη θαυματουργή δημιουργία θέσεων απασχόλησης, εδώ ή εκεί. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Και τίθεται και ένα θέμα αρχή. Εγώ δεν είμαι υπέρ των ειδικών δικαιοδοτικών συστημάτων που θα επιλύουν τις διαφορές και διαιτητικά δικαστήρια μεταξύ επενδυτών και επιχειρήσεων. Μας λέει η Επιτροπή μην ανησυχείτε, δεν αφορά μόνο τις πολυεθνικές, αφορά και τις μικρομεσαίες, αλλά για άλλη μια φορά θα είναι γνωστή συνήθεια που άλλα μας λέει και τελικά στην πράξη δεν θα ισχύει αυτό και δεν θα ωφελήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα λένε ότι θα μπορούν να υποφεληθούν, αλλά στην πράξη δεν θα αποδειχθεί αυτό και δεν υπάρχουν και εγγυήσει για τον καταναλωτή, τον πολίτη, τον εργαζόμενο στο Βιετνάμ. Και αυτό μας ενοχλεί. Αλλά, εν πάση θα γίνει συζήτηση και θα εκθέσουμε τι απόψει μα. Ευχαριστώ.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 Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή και θέλω να πω ότι εγώ ε, συμφωνώ ε, πράγματι να τα ξεχωρίσουμε αυτά, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Αυτό έγινε με τη Σιγκαπούρη, γίνεται και με το Βιετνάμ και αυτό να κάνουμε και στο μέλλον. Από την 1η Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς το εμπόριο είναι απόλυτη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν θα είναι μεικτή αρμοδιότητα. Κατά να πω ότι ε, υπήρξαν διάφορες αναταραχές και στο Βέλγιο σχετικά με τη Συμφωνία ΣΥΤΑ και γι' αυτό λοιπόν ρωτώ ποιες είναι οι πληροφορίες που παίρνει η Κομισιόν από τα κράτη-μέλη ε, σχετικά με το κατά πόσον ε, τις συμφωνίες τις εμπορικές τις εγκρίνουν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Την περίπτωση του Βιετνάμ πώς την αξιολογείτε, με ποιο βαθμό δυσκολίας. Και το τρίτο είναι θέλω να επισημάνω ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα επαγγελματικό δικαστήριο με επαγγελματίες δικαστές και για επιχειρήσεις ε, που αναλαμβάνουν κινδύνους ε, πρέπει να υπάρχουν ε, αυτά τα δικαστήρια τα οποία είναι και απόλυτα συμβατά με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει πόσο μάλλον μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και αυτά όλα δίνουν τη δυνατότητα να καταφύγει κανείς σε ένα τοπικό δικαστήριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καβατσίνη. Εγώ ε, να επανέλθω στο βασικό πρόβλημα, το οποίο το έφτιαξαν αρκετοί συνάδελφοί μου. Έχουμε ή δημιουργούμε ένα σύστημα με αυτή τη συμφωνία με το Βιετνάμ, ένα σύστημα το οποίο δημιουργεί ε, ανισορροπία ανάμεσα στους επενδυτές ε, που ζητούν κάποιες ιδιαίτερες ευκολίες, επενδυτές οι οποίοι είναι πολύ επιφυλακτική και Παράλληλα όμως ε, δεν ε, γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμετέχει σε αυτήν την, ε, τη διαπραγματεύσεις στη Γενέβη. Δεν υπάρχει ακόμα η εφαρμογή της due diligence και γι' αυτό θεωρώ ότι δημιουργούμε αυτή τη στιγμή ένα άδικο σύστημα. Ε, θέλω να τα επισημάνω αυτά τα προβλήματα. Το θέμα των δικαστηρίων προφανώς ήταν απαραίτητο να συμβεί, αλλά δεν αρκεί. Ε, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, ε, δεν αρκεί να βασιζόμαστε σε διαδικασίες. Πρέπει να ζητάμε και την τροποποίηση της νομικής βάσης. Αυτή η νομική βάση δεν μπορεί να καλύπτει βέβαια ό,τι επιθυμεί κανείς σε αυτόν τον πλανήτη. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συζήτηση για ε, γενικότερες ε, μεταρρυθμίσεις που πρέπει να λάβουν χώρα. Η κυρία Κιόνιχ. Ευχαριστώ. Κάποια σχόλια για την Συμφωνία Προστασίας των Επενδύσεων. Σωστά επισημάνθηκε πως ε, έγινε μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ώστε να ε, λάβουμε υπόψη μας και την ομοδότηση του δικαστηρίου για τη συμφωνία με τη Συγκαπούρη. και επιβεβαιώνω αυτή η συμφωνία προστασίας των επενδύσεων περιλαμβάνει πλήρως ε, το δικαίωμα ρύθμισης. Άρα και στην περίπτωση αυτή υιοθετήσαμε τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος ε, του δικαστηρίου, των, ε, των επενδυτικών δικαστηριών είναι κάτι θετικό, λαμβάνει υπόψη ε, τις ανησυχίες μας. Ένα σύστημα πλέον που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών, μεγαλύτερη διαφάνεια και τρίτα μέρη και οι των πολιτών και τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να προσφύγουν ε, σε οποιοδήποτε δικαστήριο και να καταθέσουν ε, τις ε, εκθέσεις τους. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα πέραν του ότι είναι περιορισμένο το κόστος ε, πρόσβασης ε, σε αυτή τη διαδικασία της επίλυσης επενδυτικών διαφορών από τις ΜΜΕ, υπάρχουν ε, και δυνατότητες παροχής οικονομικής υποστήριξης στις ΜΜΕ που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το σύστημα επίλυσης διαφορών. Ξεκίνησε αυτό στις συζητήσεις με, για τη Συμφωνία ΣΥΤΑ και θα ισχύει και για τη Συμφωνία εταιρική ε, σχέση ε, και συνεργασία με το Βιετνάμ. Οι ομάδες ε, τη Κοινωνία των πολιτών και οι χώρε συμβουλευτικέ ομάδε καλύπτουν όλου τους κάδους συμφωνίας και τη Συμφωνία Προστασία των Επενδύσεων. Καλύπτονται και τα δύο λοιπόν σκέλη τη συμφωνία από αυτέ τι εγχωρίε συμβουλευτικέ ομάδε για τη δέωση επιμέλεια. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πω είναι ένας τομέας ε, για τον οποίο έχουμε συζητήσει πολύ με τους Βιετναμέζου. Θέλουν και αυτοί καλές επενδύσει και όπως γνωρίζετε πράγματι θα αναλυφθούν δράσεις από την Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, δέουσα επιμέλεια, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Υπήρξαν και κάποιες ερωτήσει για την εφαρμογή, αλλά είπα ότι και η δική μα πλευρά και το Βιετνάμ εστιάζει σε αυτή ε, σε, αυτό, σε αυτή την πτυχή. διαδικασία έγκριση ε, από τα κράτη-μέλη, τελευταίο σημείο, είμαστε σε στενές επαφέ με τα κράτη-μέλη για την κύρωση και τη συμφωνία προστασία των παιδιών και τη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Όπως και με τις ΕΣ, έτσι και ε, σε αυτή την περίπτωση τις ε, συζητήσεις τις είχαμε πριν την, ε, το καλοκαίρι και θα εξαρτηθούν τα κράτη-μέλη και στις δύο περιπτώσεις. Το θέμα σχετίζεται με την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Είναι θέμα των κρατών μελών, εμείς όμως το παρακολουθούμε και όποτε και εφόσον χρειαστεί μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ κύριο Ζαχράτη. Θέλει το λόγο, όχι. Ίδια προθεσμία λοιπόν, 11 Νοεμβρίου για την κατάθεση τροπολογιών, 5 ώρα το απόγευμα. Τα ίδια ισχύουν με αυτά που είπα για το 8 και το 9. Και περνάμε ευθύ αμέσω στο σημείο 12, έτσι λίγο εντάχει βέβαια, γιατί έχουμε και την συνεδρία των συντονιστών. Νομίζω θα καθυστερήσει για 15 λεπτά περίπου. Επομένω, ερχόμαστε στο σημείο 12, χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτική Συνδρομή, στο χασιμητικό βασίλειο τη Ιορδανίας. Για δεύτερη φορά το συζητούμε. Θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στην εισηγητρία μα, την κυρία Ριτζιμέντη. E καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε, καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο που έχει επιτελέσει. Έτσι καταφέραμε και εμείς να διατυπώσουμε πρόταση ώστε να δοθεί νέα ε, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στο χασιμητικό βασίλειο της Ιορδανίας. Είχα την τιμή να μονοτεθεί ε, ο ρόλος της εισηγήτριας για το θέμα. Και ενέκυψα τις τελευταίες εβδομάδες στο θέμα αυτό και παρουσιάζω αυτήν την έκθεση. Γνωρίζετε ότι η στη Συρία είχε καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση και στο βασίλειο της Ιορδανίας με άνευ προηγουμένου ροή μεταναστών, πολύ μεγαλύτερη από άλλες χώρες, παρά το μεταναστευτικό πρόβλημα. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι η χώρα αυτή κατέβαλε πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες για να υποδεχθεί και πρόσφυγες στις αστικές της περιοχές. Και παρά τις δυσκολίες, οι εν λόγω πρόσφυγες έχουν εγγυημένη ε, δημόσια ε, και προσιτή οικονομικά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και πρόσβαση στην αγορά εργασίας ε, έτσι έλεγαν οι δεσμεύσει που είχαν αναλάβει οι Ιορδανοί. Και έτσι ε, έχουμε μια σχετικά αποδεκτή πίεση στις ε, υπηρεσίες υγείας και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. και στην παιδεία γίνονται προσπάθειες. Επίσης μεγάλη προσπάθεια γίνεται στον ε, τομέα της καταπολέμησης της, της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας και υπάρχει και εκεί έχουν εγκριθεί ad hoc νόμοι και ειδικά προγράμματα. Το βασίλειο της Ιορδανίας είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος στη Μέση Ανατολή. Προωθεί τη δημοκρατία και έχουν πάρει και μέτρα για τη βελτίωση κατάσταση των γυναικών. στην αρχή είμαστε, στα Σπάργανα. Υπάρχουν όμως και δικαστικές εξελίξεις, ε, παραδείγματος χάρη τροποποιήθηκε το, ο ποινικός κώδικας, που σήμερα μιλάμε για έναν ποινικό κώδικα ο οποίος ε, θεσπίστηκε το 2017, δεν επιτρέπει τους ε, δράστες που έχουν, κάνει, που έχουν ασκήσει βία σε βάρος γυναικών να έχουν ελαφρυντικά ή να μειωθούν οι ποινές τους. Και για μας αυτό έχει σημασία. Θέλουμε ένα σταθερό εταίρο. Χάρη στις ε, συμφωνίες των τελευταίων ετών υπάρχουν και καλύτερες συνθήκες και ευνοϊκότεροι όροι για επενδύσεις στη χώρα. Βέβαια, δεν μπορεί να βασίζεται η Ορδανία μόνο στην ε, μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση. Είναι όμως και αναμφίβολο ότι χάρη στη βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα και χάρη στην κατάλληλη πολιτική ανταπόκριση, η Ορδανία μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να παραμείνει σε σταθερή σχετικά κατάσταση και να συνεχίσει τη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Σε αυτό το πλαίσιο έδειξε η Ορδανία ότι αξίζει την μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, την επιπλέον αυτή συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό κατ' εμέ να θεσπιστούν όλα τα δέοντα συστήματα ελέγχου για να επαληθεύεται ότι γίνεται σωστή χρήση των κονδυλίων. Άρα πρέπει να επαναλάβουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη και προσιλωμένη ε, στην ε, υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλει η Ορδανία. Και ελπίζω το ψήφισμα που σας προτείνω να υπερψηφιστεί και να εγκριθεί. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό, κάθε σκιώδης εισηγητής, ένα λεπτό Χάνσεν για το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ Μπέρντ. Μιλώ εκ μέρου του κ. Ντανζάν, ο οποίο ε, ε, ταυτόχρονα πρέπει να είναι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο κ. Ντανζάν θέλει να ευχαριστήσει την εισηγήτρια κ. Ρετζιμέντη για το έργο τη και είναι ευνοϊκά δικημένο απέναντι στην πρόταση για χορήγηση νέα μικροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία για να στηριχθεί η Ιορδανική οικονομία που είναι σε έφραυστη κατάσταση, επειδή χρειάζονται εξωτερική χρηματοδότηση και υπάρχουν και κάποιε αδυναμίε σε αυτή τη χώρα. Ο κ. Νασάν θέλει να υπογραμμίσει ότι είναι στρατηγικό εταίρο, σημαντικό εταίρο τη Ένωση η Ορδανία, ιδίω λόγω του σημαντικού ρόλου που έχει στην προώθηση σταθερότητα και τη ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Η συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και όλων των διεθνών εταίρων είναι κάτι απαραίτητο και ευκταίο. Αυτό το πρόγραμμα είναι θετικό δείγμα και μήνυμα που στέλνει η Ένωση στις χώρες της περιοχής ότι θέλει να βοηθήσει δηλαδή ε, τις χώρες, η Ένωση που θέλουν να ε, προβούν σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Σάντος, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να πω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή. Ξέρουμε ότι το βασίλειο της Ιορδανίας είναι πολύ σημαντικός εταίρος στην ε, περιοχή ε, αυτή. Αυτή τη στιγμή υφίσταται πολύ μεγάλη πίεση, έχει υποφέρει πολύ διότι είναι πολύ κοντά στην κρίση της Συρίας και έχει υπάρχει μεγάλη ροή ε, προσφύγων στη χώρα. Πρόσφυγες τους οποίους έχει υποδεχθεί το βασίλειο της ε, Ιορδανίας, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, υιοθετούν πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις όχι μόνο στο, στην εσωτερική του νομοθεσία, αλλά κάνουν τα απαραίτητα βήματα για τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, έτσι ώστε να είναι μια κοινωνία όλο και πιο ανοιχτή. Έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή. Σε αυτή τη συμφωνία τώρα διάφορες δεσμεύσεις είναι αυτές που έχουν υιοθετήσει. για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη μακροοικονομική βοήθεια. Σε κάθε περίπτωση στηρίζω πλήρως αυτά που προτάθηκαν. Και πιστεύω ακρατάντος ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε αυτό το ισχυρό μήνυμα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να βοηθήσει να σταθεροποιήσει αυτή τη χώρα και μέσω αυτής και την υπόλοιπη περιοχή. Πρέπει να προάγουμε αυτές τις πολύ σημαντικές αξίες που είναι η ανάπτυξη και η δημοκρατία. Είναι πολύ σοβαρή η αταλάντευτη προσήλωσή μας στα ανθρώπινα, στα δικαιώματα. Αυτό πρέπει να συνεχίσει να πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην παραιτηθούμε ποτέ από αυτό το στόχο. Και αυτό φαίνεται πολύ καλά από τα συμπεράσματα του εισηγητή. Ο από το Ρινιού παρακαλώ επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Ως και όδης εισηγητής για το Ρινιού θέλω να εκφράσω την στήριξή μου στη χορήγηση αυτής της μακροοικονομικής βοήθειας στο Βασίλειο της Ιορδανίας η οποία θα συμβάλλει, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, τη στήριξη του βασιλείου της Ιορδανίας εν ώψη και λόγω της μεγάλης κρίσης στη Συρία. Παρ' όλα αυτά μας φαίνεται σημαντικό αυτή η σημαντική οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έρχεται για τρίτη φορά να ε, συνδέεται με, κάποιες, ε, με την υλοποίηση ορισμένων δεσμεύσεων της κυβέρνησης που έχει αναλάβει κατά προτεραιότητα. Βελτίωση του συστήματος πόσιμου ύδατος, βελτίωση του ηλεκτρικού συστήματος και βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας. Ζητούμε αυστηρή εποπτεία και παρακολούθηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης των δράσεων και μεταρρυθμίσεων που ε, υιοθετεί η Ορδανία μετά την απόκτηση, μετά τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Βοήθειας και να τηρείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενήμερο. Επομένως στηρίζουμε ανεπιφύλακτα την οικονομική βοήθεια, ωστόσο Επιτρέψτε μου να κάνω μία μικρή παρατήρηση, γιατί η ομάδα ID που έχει αναλάβει την έκθεση αυτή ε, έχει κάποιες αντιφατικές ιδέες. Πολλά από τα μέλη του ID πηγαίνουν στη Συρία και στηρίζουν τον Μπασάρα Λασάντ και είναι ως φιοκάμπτες αυτού και από την άλλη έρχονται και στηρίζουν ε, την Ιορδανία εδώ είναι αντίφαση αυτό. Επομένως, ε, ε, αυτή η πολιτική ομάδα ε, ποτέ δεν χάνει ευκαιρία να μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε και να εντοπίσουμε τις αντιφάσεις μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φράγκος δεν είναι εδώ, γι' αυτό και θα δώσω το λόγο στον κύριο Μορέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζουμε καλά στην Επιτροπή μας. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία το έχουμε συζητήσει επισταμένως και εγώ έχω μεταβεί στην Ιορδανία και έχω συζητήσει με τις αρμόδιες αρχές και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή στην πράξη. Ναι, είναι σημαντική η εταιρική σχέση, δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, αποσταθεροποιήθηκε βία η χώρα αυτή από αυτά που έγιναν στις Συρία και ε, βέβαια για θέματα υποδοχής προσφύγων τα νούμερά τους είναι αστρονομικά. Δεν είναι αυτό που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη να αντιμετωπίσουμε. Το Ιορδανικό κράτος δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να υποδεχθεί όλους αυτούς τους πρόσφυγες. Εγώ είμαι πάντοτε υπέρ της οικονομικής βοήθειας. Αυτό το οποίο με ενοχλεί όμως είναι το εξή. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να επιβάλλουμε σε μια χώρα σαν την Ιορδανία, η οποία έχει αποδυναμωθεί ιδιαίτερος. Τι κάνουμε, τους λέμε ορίστε να η οικονομική βοήθεια και να οι τι γίνεται όμω με τι δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει. Το ίδιο συμβαίνει και με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Όταν έχουμε νεοφιλελεύθερη ατζέντα και θέλουμε να κάνουμε μια χώρα να την υιοθετήσει και την επιβάλλει στο λαό τη. Το έχουμε κάνει και με την Τινησία και αλλού. Χωρί να λάβουμε υπόψη τι μπορεί να κάνει αυτό ο λαό και τι είναι καλό ε, για αυτό το λαό, ε, τότε ε, οδηγόμαστε, οδηγούμαστε σε καταστροφή. Το λογικό είναι να ακυρώσουμε τα χρέη ή να κάνουμε κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν είναι σωστή η πολιτική που υιοθετείται αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να το σκεφτούμε για το μέλλον, για τη μελλοντική μας προσέγγιση. Γιατί του ζητούμε πράγματα που δεν είναι εφικτό να πράξουν. Ο πρέσβης της Ιορδανία, παρακαλώ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νόμιζα ότι είχα τέσσερα λεπτά στη διάθεσή μου, αλλά δεν πειράζει. Όλοι είπαν κάτι για την Ιορδανία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές που αναφέρθηκαν στη χώρα μου, τους συναδέλφους τους, ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όντως μεταφέρατε την ευρύτερη εικόνα που επικρατεί στη χώρα. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου να σας δώσω κάποια στοιχεία για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, στην πράξη, στην Ιορδανία. Είμαστε στο προσκήνιο, στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης της Παστικοποίηση και τη τρομοκρατία. Εμεί είμαστε πολύ αξιόπιστος εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνεργασία για την καταπολέμηση τη τρομοκρατίας, την καταπολέμηση των ξένων μαχητών, την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων για όλα αυτά. Είμαστε ο καλύτερος συνεργάτης Ευρωπαϊκή Ένωση. και με περηφάνεια σα λέω ότι η χώρα μου διαδραμάτισε ρόλο κλειδί για την ακύρωση ε, τρομοκρατικών σχεδίων που κατεργάζονταν και επεξεργάζονταν τρομοκράτε που επρόκειτο να πλήξουν ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε. Τα εξουδετερώσαμε τα σχέδια αυτά με καθοριστική συμβολή τη ε, Ιορδανία. 3,6 εκατομμύρια πρόσφυγε βρίσκονται στη Συρία από 52 διαφορετικέ ε, εθνικότητε, από τη Συρία, από το Ιράκ, την Ιεμένη, την Παλαιστίνη βεβαίω, του Παλαιστινίου και ε, Σύρου επίση. 10 εκατομμύρια είναι ο πληθυσμός της Ιορδανία, ο εγχώριος πληθυσμός, 6,5 εκατομμύρια είναι οι γηγενείς Ιορδανοί και 3,5 εκατομμύρια οι πρόσφυγες. Μοιραζόμαστε τους σπάνιους πόρους της Ιορδανίας σε ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα ηλεκτρισμού ενέργειας και τους υδάτινους πόρους οι οποίοι λείπουν, ε, στους οποίους υστερούμε. Κατά 90% ζουν σε κοινότητες υποδοχής και κατά 10% σε καταβλισμούς. Όλη η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνει στους καταβλισμούς. Το 90% όμως των προσφύγων ζουν στα αστικά κέντρα και μοιράζονται τους πόρους με την υπόλοιπη αστική κοινότητα. Και πρέπει να διορθωθεί αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει βοήθεια μόνο στους καταβλισμούς, γιατί 10% μόνο μένουν σε καταβλισμούς σε εμάς. Παρά τις προκλήσεις που έχουν υψωθεί για την Ιορδανική οικονομία, ε, τελικά είχαμε πολύ υψηλή ανεργία, 19,2% το 2019, 40% ανεργία των νέων. Ε, βλέπετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης έχουν καταλάβει οι Σύριοι και τους έχουν, τις έχουν πάρει από τους Ιορδανούς. Παραμένουμε όμως ανεκτική σαν Συνεχίζουμε να έχουμε θετικό βλέμμα έναντι των Σύρων προσφύγων εμείς οι Ιορδανοί. 1,4 δις ευρώ. Είναι μικρό το νούμερο στα μάτια σας, αλλά για μια χώρα σαν την Ιορδανία με πολύ φτωχή οικονομία είναι τεράστιο το νούμερο αυτό. Το κόστος υποδοχής των προσφύγων και ο αντίκτυπος που έχουν από την αρχή της κρίσης μέχρι τα τέλη του 2018 ανήλθε στα 11 δις ευρώ σχεδόν. Είναι τεράστιο το νούμερο για μια χώρα σαν τη δική μας, για μια οικονομία σαν τη δική μας. Ο έμεσος, έμεσος αντίκτυπος της κρίσης της Συρίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του UNDP, του αναπτυξιακού προγράμματο των Εθνών είναι, σύμφωνα με τις αναλύσεις, ο ως αντίκτυπο ανέρχεται σε περίπου σχεδόν 3 δις ευρώ ετησίως. Είναι το κόστος υποδοχής των προσφύγων για τη δική μας χώρα με βάση τις μελέτες του ΟΗΕ και του προγράμματος για την αναπτυξιακή βοήθεια. Για να παραμείνουν οι Σύροι κοντά στα σπίτια τους στην Ιορδανία, θυμάστε την κρίση του 2015 και πόσο υπήρχε ο κίνδυνος επέκτασης της στις ευρύτερες γειτονικές περιοχές, προσπαθούμε να τους στεγάσουμε κοντά στα σπίτια τους, να τους δώσουμε ελπίδα, να δώσουμε τις υπηρεσίες τις κρατικές να μπορούν να υποφεληθούν από αυτές Επιτρέψαμε στους Σύρους πρόσφαγες εντός των καταβλισμών να έχουν άδειε εργασίες, άδεια και να εργάζονται και εκτός καταβλισμών. Η κυβέρνηση έδωσε άδειε εργασίες για το κατασκευαστικό κλάδο, για την ελεύθερη μετακίνησή τους, για ιατρικά πιστοποιητικά και ούτω καθεξής ελεύθερα και τα προνόμια και οι υπηρεσίε που τους δίνουμε είναι πάρα πολλά. Και ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, για να διευκολύνουμε τους Σύρους πρόσφυγες, η κυβέρνηση ε, δέχθηκε να εγγραφούν στα σχολεία και στις σχολές. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλ, ε, εκπαίδευση δημόσια δωρεάν. Ε, ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Τα παιδιά που έχουν γραφτεί στα δημόσια σχολεία είναι περίπου 140.000. 140.000 παιδιά από τη Συρία φοιτούν στο δημόσιο σχολείο της Ιορδανίας, το οποίο δουλεύει με διπλοβάρτια. Ε, σε ορισμένα σχολεία έχουμε τριπλές βάρδιες για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε τους σύρους μαθητές. Έχουμε ανοίξει όλες τις ιατρικές υπηρεσίες. Ε, η ίδια πρόσβαση στην περίθαλψη έχουν όπως έχουν οι Ορδανοί πολίτες. Και θα σταματήσω κάπου εδώ γιατί όλοι μίλησατε πολύ θετικά για την Ορδανία. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να παρουσιάσω τα τεκτενόμενα στη χώρα μου. Ε, όσον αφορά τους και οδησυγητές. δυστυχώ ξέχασα τους ε, πράσινου. Φυσικά ε, θέλουμε να διατηρηθεί η χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία. Υπάρχουν πολλέ ε, που πρέπει να αντιμετωπίσει η χώρα, ιδίω ό,τι αφορά την κατάσταση των προσφύγων. Όμω, έχουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Όπω είπαν κάποιοι συνάλληλοι, δεν θα πρέπει να εστιάζουμε μόνο στα οικονομικά στοιχεία των ε, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και στο κράτο δικαίου. Δράτω με τις ευκαιρίε επίσης για να πω ότι υπάρχει μια ασυνέπεια στι πολιτικέ τη Ένωση, ε, όταν μιλάμε για μη διαχείριση ε, του μεταναστευτικού από τη μία και από την άλλη οθέτηση προγραμμάτων που ουσιαστικά εκχωρούν σε τρίτε χώρε καθήκοντα που οι ίδιες δεν ε, φέρουν σε πέρας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Εκ μέρους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γκρασία, για δύο λεπτά. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Ρετζιμέντη Και πρέπει να σας πω ότι εμείς ε, ε, στηριχθήκαμε, ενθαρρυνθήκαμε πάρα πολύ από την ταχύτητα με την οποία προχωράει αυτή η έκθεση. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας στο Συμβούλιο κατά τις επόμενες εβδομάδες μέχρι να εγκριθεί η εισήγηση. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η Ορδανία εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις. Προφανώς και έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, αλλά ακόμα υπολείπονται αρκετά. Ε, Πράγματι, η, βοήθεια, η μακροοικονομική θα μπορούσε να βοηθήσει για να επιτευχθεί πρόοδος. Ε, κάποια σχόλια που λέξαν σήμερα αφορούν την αιρεσιμότητα. Ε, στην περίπτωση αυτή η Ορδανία πρέπει να οικειοποιηθεί τις μεταρρυθμίσεις. Ε, υπάρχουν ακόμα προβλήματα στις μεταρρυθμίσεις και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό μάθημα που έχουμε εξάγει από την εμπειρία μας και από προηγούμενες περιπτώσεις όπου χορηγήθηκε μακροοικονομική βοήθεια. Αναφέρθηκαν θέματα όπως το επιχειρηματικό περιβάλλον, ε, ίδρυυση, ηλεκτρισμός, ε, φορολογία. Αυτά είναι θέματα που αφορούν ε, το ενδεχόμενο της ερεσιμότητας σε σχέση με την μακροοικονομική χρηματοδότηση. Τέλος, όσον αφορά την χρήση των κονδυλίων, έχουμε την, το μνημόνιο συμφωνίας, ε, τη συμφωνίες συνεργασίας. Εκεί περιλαμβάνεται και μία ρήτρα για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να τηρηθεί. Και Αυτά όλα σημαίνουν ότι τα κονδύλια και η βοήθεια χορηγείται γενικότερα, όχι για συγκεκριμένους σκοπούς. Πάντως είναι πολύ σημαντικό τα κονδύλια να τύχουν σωστή διαχείρισης και να υπάρχει και λογοδοσία στον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισηγήτρια παρακαλώ. Ε, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Νομίζω ότι το θέμα εξετάστηκε ικανοποιητικά και δεν νομίζω ότι ζήτησε κανείς ε, κάποια περαιτέρω διευκρίνηση. Ως εκ τούτου και εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Πολύ ωραία. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 14η Νοεμβρίου για κατάσταση απολογιών. Είναι μέρα των γενεθλίων μου μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Και θα ψηφίσουμε στην ΙΝΤΑ στις 13 Δεκεμβρίου. Ε, θα κάνουμε ε, διάλειμμα πολύ σύντομο για ένα λεπτό και μετά θα έχουμε συνεδρίες των συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Παρακαλώ.